Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτο στοιχείο τη ε, τη διάταξης είναι το θέμα της χρηματοδότησης καινοτομία σε παγκοσμό και ευρωπαϊκό επίπεδο με εισηγήτρια την ανυπόδηματά, στην οποία δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο εισαγωγικά. Είναι η τελευταία μας συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η έκθεση για τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης έχει μια σημαντική προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρέπει να διερευνήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις εναλλακτικέ λύσεις για νέες πηγές και πόρους χρηματοδότησης σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και οι εθνικοί προϋπολογισμοί, τα κράτη-μέλη, το έχουν περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ. Αυτή είναι μια διάσταση, σημαντική διάσταση των καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης. Η άλλη σημαντική διάσταση είναι ο ρυθμιστικός ρόλος των μέσων αυτών, ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν τόσο το πακέτο της ε, χρηματοπιστωτικής εποπτείας και ρύθμισης, όσο και το πλαίσιο της ε, νέας οικονομικής ε, διακυβέρνησης και φυσικά της στρατηγικής ΕΕ 2020. Και φυσικά ε, η στροφή στα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης πιστεύω ότι αποτελεί και μία ευκαιρία για το Κοινοβούλιο για να αναδείξει ακόμα μία φορά την κοινοτική προσέγγιση, την ενωσιακή προσέγγιση έναντι της διακυβερνητικής, δίνοντας και ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, μπορούμε να προωθήσουμε λύσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν χωρίς να υποκαθιστούν τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο εθνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, για να παραπέμψω και στην ε, χθεσινή μας συζήτηση, τα καινοτόμα στη χθεσινή μας συζήτηση για το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης, τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως κίνητρο, ως καρότο που λέγαμε και χθε, εξισορροπώντας τη λογική των ποινών και των κυρώσεων και άρα να συμβάλλουν ώστε οι πολιτικές της Ένωσης να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές. Έρχομαι στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, οι οποίες έχουμε καταλήξει μετά από 1,5 ε, μήνα διαπραγματεύσεων και σειρά συναντήσεων με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Θέλω να θυμίσω ότι κατατέθηκαν 200 τροπολογίες και ότι είχαμε σημαντική διάσταση απόψεων σε ορισμένα σημεία κλειδιά Οπότε έπρεπε να βρούμε κοινό έδαφος για να καταλήξουμε σε ένα συνεκτικό κείμενο που θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ε, αποδοχή ώστε να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εκφραστεί με μια ενιαία φωνή και να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή στο θέμα αυτό. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ε, που έχουμε επεξεργαστεί ακολουθούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της ε, έκθεσης. Ο πρώτος πυλώνας αφορά, όπως ξέρετε, την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Θα πω πού έχουμε συμφωνήσει και τι εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρεμότητα. Έχουμε καταλήξει λοιπόν σε συμφωνία σχετικά με τις σημαντικές δυνατότητες, τώρα αναφέρομαι στην συμβαστική τροπολογία στην παράγραφο 5 του κειμένου, ε, που αφορά στις σημαντικές δυνατότητες για επιπρόσθετα έσοδα, επιπρόσθετους πόρους, ε, από ένα φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τις μέχρι σήμερα εξελίξεις στο επίπεδο του G20 και την ε, ανάγκη που αποδεχόμαστε όλοι να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση μιας παγκόσμιας συμφωνίας στο θέμα αυτό. Ε, στην ανάγκη να πάρουμε τα σωστά μαθήματα από νομοθεσίες αντίστοιχες παρεμφερείς ε, και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα κράτη-μέλη το προηγούμενο διάστημα, την πεποίθηση ότι αν και η υιοθέτηση ενός ε, φόρου ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσε να έχει κάποιες αρνητικές συνέπειες ως προς τη μετανάστευση κάποιων συναλλαγών προς άλλες δικαιοδοσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα θα συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της ε, διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στο χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα. Τις, ε, έχουμε συμφωνήσει στις τεχνικές, τεχνικές πτυχές σχετικά με την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ειδικότερα στην προστιθέμενη αξία των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, οι οποίοι καθιστούν πολύ πιο εύκολη την εισαγωγή στο τεχνικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μελέτη επιπτώσεων, η οποία θα λαμβάνει υπόψη πτυχές όπως η γεωγραφική ασυμμετρία, η δυνατότητα διαφοροποιημένων συντελεστών, το ποιος θα αναλαμβάνει τελικά το κόστος της, ε, της φορολόγησης, το φορολογικό βάρος, το πεδίο εφαρμογής και τέλος τη διαχείριση των εσόδων, τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις για τη διαχείριση των εσόδων από τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ε, δύο είναι τα σημεία τα οποία έχουμε αφήσει ε, ανοιχτά. Ε, ξεκινώ από την παράγραφο 1, όπου κάνουμε αναφορά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του περασμένου Μαρτίου για μελέτη επιπτώσεων σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από την τελευταία συνάντηση με τους Σκιώδης την περασμένη Τετάρτη στο Στρασβούργο, ε, είχαμε μια πρόταση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο θέμα αυτό ε, που παραπέμπει και σε άλλες παραγράφους του ψηφίσματος της, ε, της 10ης Μαρτίου του 2010 και προτείνει προκειμένου να υπάρξει διέξοδος και να μπορέσουμε να βρούμε κοινό έδαφος να χρησιμοποιήσουμε τον όρο φόρη στο χρηματοπιστωτικό ε, τομέα, φόροι χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, και αυτή είναι μια διατύπωση που θα μπορούσε ε, να γίνει αποδεκτή εάν πρόκειται να διευκολύνει την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Η εκκρεμότητα παραμένει στην παράγραφο 7 του κειμένου, όπου μετά από μια σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων καταλήξαμε να προτείνουμε ως συμβιβαστική ε, τροπολογία το κείμενο της παραγράφου 73 της ε, έκθεσης Επιτροπής για την κρίση, της έκθεσης ε, Μπέρες. Είναι λέξη προς λέξη η παράγραφος αυτή, στην παράγρα... η παράγραφος 73 της έκθεσης Μπέρες, στην παράγραφο 7 του, κειμένου του δικού μας. πρόκειται, θυμίζω, για το κείμενο που υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Και θυμίζω ότι ε, με την παράγρα... η παράγραφος εκείνη αναφέρεται στην επίτευξη συμφωνίας για φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και αν αυτό δεν καταστεί ε, δυνατόν ε, σε πρώτη φάση, ως πρώτο βήμα να γίνει αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά σε ό,τι αφορά την, τον, το κεφάλαιο που αφορά τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, το κεφάλαιο που αφορά τα ε, ευρωομόλογα και τα επενδυτικά ε, ευρωομόλογα. Ε, καταρχήν έχουμε καταλήξει σε ένα νέο τίτλο για να καταστήσουμε πιο ξεκάθαρη την διάκριση ανάμεσα στα ευρωομόλογα χρέους και στα επενδυτικά ευρωομόλογα. Στην πρώτη περίπτωση η συμβιβαστική τροπολογία ε, στην οποία ε, νομίζω ότι καταλήξαμε στην τελευταία μας συνάντηση, ε, κάνει μία επισήμανση στο γεγονός ότι υπάρχει σήμερα μία σημαντική συζήτηση ως προς το θέμα αυτό, μία σημαντική συζήτηση δηλαδή ως προς την χρήση των ευρωομολόγων ως εργαλείου κοινή διαχείρισης μέρους του χρέους. Σημειώνει ότι έχουν κατατεθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες και προτάσεις γύρω από το θέμα αυτό τον τελευταίο καιρό και ε, τέλος παραθέτει το απόσπασμα από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήσαμε στις 16 ε, Δεκεμβρίου για το μόνιμο ε, μηχανισμό σταθερότητας όπου με βάση το ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει ένα ξεκάθαρο πολιτικό σήμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διερεύνηση της σκοπιμότητας της έκδοσης ευρωομολόγων. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ομόλογα επενδύσεων, τα ευρωομόλογα επενδύσεων, η συμβιβαστική τροπολογία ε, τάσεται υπέρ της έκδοσής τους για τη στήριξη της ανάπτυξης, των επενδύσεων και τη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων ΕΕ2020. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο που αφορά την ε, φορολογία στον τομέα της ενέργειας, έχουμε και εκεί καταλήξει αρκετά νωρί σε πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, τις αναφέρω εντάχει. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, που θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στη φορολογία στον ε, τομέα της ενέργειας και η ανάγκη για ε, μετάβαση του φορολογικού άκθους από τομείς όπως η εργασία σε τομείς που προκαλούν περιβαλλοντική μόλυνση. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο βεβαίως αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία στον τομέα της ενέργειας που ξέρουμε ότι επίκειται ε, ζητάμε στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης να περιλαμβάνονται τα κριτήρια της εκπομπής ρήπων διοξιδίου του άνθρακα και το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας, το διπλό όφελος της, ε, της φορολογίας άνθρακα σε ό,τι αφορά την, ε, τη συμβολή μιας τέτοιας φορολογίας στην αλλαγή συμπεριφοράς, την ανάγκη για μια διεθνή συμφωνία καταρχήν για φορολογία άνθρακα στο πλαίσιο του G20 και την εναλλακτική του, Border Tax uh, Adjustment στο επίπεδο του WTO, την προοπτική για ένα φόρο αξίας με βάση τον άνθρακα στο πρότυπο του φόρου προστιθέμενης αξίας. Και φυσικά θέλω να θυμίσω ότι στον τομέα αυτό θα έχουμε και τις ε, προτάσεις ε, που, από την ε, Επιτροπή Έρευνας, Ενέργειας και Βιομηχανίας, την Επιτροπή Ήτρε. Τέλος, ό,τι αφορά το θέμα των καινοτόμων μέσων για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών πολιτικών, καταλήξαμε σε μια συνολική συμβιβαστική πρόταση, ωστόσο και εκεί θα έχουμε την ε, σημαντική συμβολή των προτάσεων της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα. Ήθελα ε, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά με την ευκαιρία του σκιώδης εισηγητές για την συνεργασία τους και για την συμβολή τους και να εκφράσω την ελπίδα να αρθεί και η τελευταία δυσκολία στην παράγραφο 7 ώστε να πάμε σε έναν καλό συμβιβασμό σε ένα θέμα που όπως είπα από την αρχή μπορούμε και πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, τολμηροί και να βρούμε λύσεις που θα προωθούν το κοινό ε, ευρωπαϊκό συμφέρον διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς για την Ευρώπη την συνοχή και την ε, αξιοπιστία του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα συμπεφωνημένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Απόδηματά. Μιλήσατε πάρα πολύ σαφώς και τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κυρία Χίμπνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι το να λάβουμε υπόψη τη δυσκολία και το ευαίσθητο αυτών των ζητημάτων είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά μεταξύ της εισηγήτριας και των σκιωδών εισηγητών για τα θέματα αυτά σε, στην κατεύθυνση ενός συμβιβασμού, αλλά όπως είπε και η κυρία Ποδηματά, έχουμε ακόμα να διατρέξουμε δρόμο για να κλείσουμε την διαπραγμάτευση και το, τη συμβαστική λύση για αυτή την πρόταση. Θα ήταν λοιπόν πρέπει και ορθό από πολιτική άποψη να μπορέσουμε να βρούμε μια τέτοια κοινή θέση και ελπίζω θα μπορέσουμε να το κάνουμε εν καιρό πριν από την ψηφοφορία της επόμενη εβδομάδα. Δεν θέλω να επαναλάβω τώρα αυτά που είπαμε στο παρελθόν. <clears throat> Απλώς θέλω να σταθώ σε μία ή δύο διαφορές που εξακολουθούμε να έχουμε υποσυζήτηση μεταξύ μας. Και όπως καταλαβαίνετε και από αυτά που είπε και η κυρία Πόδηματά, <clears throat> το πιο σημαντικό είναι ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Γιατί η πρόθεση της εισηγήτριας είναι να παραμείνει πιστή στο κείμενο το οποίο ψηφίστηκε ως έκθεση Μπερές με την βασική αυτή ιδέα να υπάρξει φόρος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και εκεί τονίζεται ότι αυτό είναι μια εφικτή επιλογή. Γνωρίζουμε όλοι και τα δυνητικά πλεονεκτήματα αλλά και τα δυνητικά μειονεκτήματα της επιβολής ενός τέτοιου φόρου μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να περιμένουμε και την έκθεση αντικτύπου και θα πρέπει να εξετάσουμε το πρόβλημα αυτό με τον πιο προσεκτικό δυνατό τρόπο. Πρέπει αυτή η διαδικασία να περατωθεί μέχρι το καλοκαίρι φέτος και αν περατωθεί αυτή η έκθεση αντικτύπου θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά μόνο έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για την αναζήτηση <clears throat> μιας κοινή συμβαστική πρότασης. Συμφωνώ με την Άννη ότι για την παράγραφο 1 όπου γίνεται η μνήα του ψηφίσματος του Μαρτίου 2010 νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση για να χρησιμοποιήσουμε τη διατύπωση που υπήρχε στο ψήφισμα όπως ψηφίστηκε πέρσι. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, για τα ευρωομόλογα και την φορολογία του άνθρακος έχουμε βρει μια συμφωνία και είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική λύση σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση των φυσικών πόρων των πόρων οι οποίοι θα προέλθουν από τη φορολογία χρηματοοικονομικών συναλλαγών δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να κόψουμε το νήμα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε και τα προβλήματα τα οποία παραμένουν πριν από την ψηφοφορία που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Ο κύριος Σμίθ έχει το λόγο τώρα. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και να συγχαρώ την κυρία Ποδηματά όπως ξέρουμε, το θέμα αυτό το αντιμετώπισε και ήταν το Χίμπνερ, πολύ δύσκολο και το ξέρουμε. Τώρα όμως το συζητάμε αρκετές ώρες και τουλάχιστον από τη δικιά μας την πλευρά των φιλελευθέρων καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τα δύο προβλήματα βεβαίως είναι πρώτα απ' όλα το FTT, ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών και τα ευρωομόλογα αλλά τα ευρωομόλογα νομίζω θα λυθούν πιο εύκολα και έχουμε νομίζω ένα κοινό κείμενο που συμφωνήσαμε πέρσι. Για το φόρο όμως θα πω πως όπως και η κυρία Χιούμπνερ ε, και το κείμενο της έκθεσης ήταν ένας δύσκολος συμβιβασμός και δεν ε, ε, μας διευκόλυναν και οι πράσινοι στο να καταθέσουμε μια προφορική τροπολογία στο τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς στο τέλος αποδεχτήκαμε το κείμενο ολόκληρο παρά το ότι είχαμε καταψηφίσει το μέρος που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι το, το πρώτο βήμα. Παρά το ότι αυτό λοιπόν ήταν στο κείμενο, τελικά υπερψηφίσαμε την έκθεση Μπερές. Και θεωρώ πως η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθεί και αυτή τη φορά. Και νομίζω πως αυτό ήταν ο, ο συμβιβασμός που επιτύχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει από την πλευρά του ΕΛΚ. Γιατί νομίζω πως ε, πρέπει και εμείς στην ομάδα μας ε, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή θα στηρίξουμε την έκθεση αν έχει αυτό το κείμενο. Αλλιώ δύσκολα θα πείσω κάποιου σύναδελφού μου που δεν είναι και τόσο υπέρ του πρώτου αυτού ευρωπαϊκού βήματος. Οπότε, κατά την απόψή μας, αυτό είναι το, το πρόβλημα που, παραμένει. Αλλά στα υπόλοιπα νομίζω έχουμε φτάσει σε συμβιβασμούς και Ολοκληρώνοντας, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χούμπνερ θέλει να επανέλθει. Θέλετε να διευκρινίσετε κάποιο σημείο. Αυτό που ανέφερε ο κύριος ε, Σμιτ. Προσπαθούσα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σαφής. Εδώ πέρα έχουμε διαφωνίες, οπότε δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δεχτούμε. Μία εβδομάδα δηλαδή πριν την τελική προθεσμία, να δεχτούμε τη διατύπωση που προέρχεται κατευθείαν από την έκθεση την περσινή που λέει σαφώς ως θεωρεί πως η εισαγωγή ενός φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν ευρύτερη και αν δεν γίνει αυτό που... Ε, γιατί νομίζω πως ε, είχαμε συνοηθεί πως θέλαμε ένα παγκόσμιο φόρο ή αν δεν είναι δυνατόν αυτό θα πρέπει να γίνει ως πρώτο βήμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε πεπισμένοι πως δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο άμεση. Πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έχουμε ακούσει τουλάχιστον τρεις φορές εδώ πέρα πώς θα οριστικοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι. Οπότε θεωρούμε πως μόνο εάν το θεωρήσει σωστό η Κομισιόν ε, μπορεί να επιβληθεί αυτός ο φόρος στο επίπεδο της Ένωσης εάν απορριφθεί από άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα δούμε τι θα γίνει με το φόρο αυτό. Αλλά χωρίς την αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, δεν μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή πλήρως τη σχέση μεταξύ πλέον εκτιμάτων και μειονεκτημάτων ενός τέτοιου φόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τη διευκρίνηση. Νομίζω πως έχουμε κάποιες μέρες ακόμα για να οριστικοποιήσουμε το κείμενο. Αυτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πότε προβλέπετε να δώσετε στη δημοσιότητα, να μας δώσετε μάλλον το έγγραφο το οποίο ανέφερε η κυρία Χιούμπνερ. Ρωτάω την Κομισιόν, λέει ο κύριος ε, Μαργάιο, πότε θα μας διαβιβάσει η Κομισιόν το έγγραφο το οποίο αναφέρατε, δηλαδή την έκθεση αντικτύπου. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα από αυτά που είπε ο κύριος Επίτροπος πριν από δύο εβδομάδες. Θα είναι έτοιμη μέχρι το καλοκαίρι η έκθεση αντικτύπου, αλλά θα μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Φίλιπ Λαμπέρ έχει το λόγο τώρα. Δεν θα ήθελα να παρευληθώ στη συζήτηση μεταξύ των ελεύθερων και του ΕΛΚ. Θέλω να πω εξή. Πρώτον, εκτιμώ την ειλικρίνεια και της Ντανούτα και όλων των άλλων στη συζήτηση. Καλή προσπάθεια, αλλά θέλω να είμαι και εγώ εξίσου ειλικρινής. Έχει σχέση με τη χθεσινή συζήτηση για τη δημοσιονομική εποπτεία και διακυβέρνηση. Μίλησα και με τους και με το ΕΛΚ και βλέπω ότι και οι δύο ομάδες επιμένουν να έχουμε μια σύγκληση προς βιώσια, βιώσιμα δημόσια οικονομικά με περικοπή των περικοπών και γρήγορη μείωση του χρέους. Είπατε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συμφωνώ. Επίσης οι ομάδες σας λένε πρέπει να επενδύσουμε στους στόχους του 2020. Ένα τμήμα είναι ιδιωτικές επενδύσεις, ένα τμήμα είναι δημόσιες. Κάθε φορά που συζητάμε πόρους που θα επέτρεπαν επενδύσεις στους στόχους 2020 για κάθε θέμα όσον αφορά τα κονδύλια η απάντησή σας είναι είτε όχι είτε θα το σκεφτούμε ή πρέπει να γίνει μια μελέτη αξιολόγησης πραγματικά παραξενεύομαι πώς συνδυάζεται πρώτα από μια μεριά το να θέλετε λιτότητα και από την άλλη επιλογή για επενδύσεις για το 2020. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί η εξίσωση αυτή, που κατά γνώμη μου δεν γίνεται, είναι αν δεν φορολογήσουμε τις επιχειρήσεις. Δεν το θέλετε. Να μην ε, φορολογήσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα. Χρειαζόμαστε μελέτη. Δεν θέλουμε την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής, γιατί η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι το πιο σωστό μέσο τότε το μόνο έσοδο που μένει είναι η φορολόγηση του εισοδήματος. Εισόδημα εργασίας, που σημαίνει και πάλι να φορολογήσουμε αυτούς που είναι οι ασθενέστεροι. Και είτε τους φορολογούμε βέβαια είτε τους ε, δίνουμε λιγότερη κοινωνική υποστήριξη, επιδόματα κλπ. Θα προτιμούσα κάποια στιγμή να μου δοθεί ευκαιρία να καταλάβω πώς βλέπετε εσείς την εξίσωση. Γιατί επαναλαμβάνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Προτείνω λοιπόν να μείνουμε στη διατύπωση της έκθεσης Μπερένς και αν αυτό είναι δύσκολο, προτείνετε να μας προτείνετε εσείς φερέγγες αναλλακτικές λύσεις. Γιατί μέχρι σήμερα λέτε περικοπή των δαπανών και όχι επιπλέον έσοδα. Αυτό λέτε. Αν το στείλουμε το μήνυμα αυτό στους πολίτες, τι να πω, δεν στέκεται. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον Φιλίπ Ιβο Στρέτζεκ. Αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα συνεχίσω στην εύγλωτη επιχειρηματολογία του κυρίου Άλμπερντς. Μερικές από τις ιδέες του είναι ενδιαφέρουσες. Εγώ όμως θα ξαναγυρίσω στην έκθεση της κυρίας Ποδηματά και εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά της γιατί το θέμα είναι περίπλοκο και όπως είπε ο κύριος Λάμπερτ είναι δύσκολο να γίνει δεκτό από μερικά κράτη-μέλη της Ένωσης. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που έχω πει για τη λεγόμενη εναλλακτική χρηματοδότηση. Είμαστε μόλις στην αρχή μιας εποχής δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη-μέλη. Η γνώμη μου και η γνώμη του, της ομάδας μου είναι ότι αυτό θα πρέπει να αντακατοπτρίζεται και στο Ευρωκοινοβούλιο. Μοιραία θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν φράσεις που να αναφέρονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι στις και επίσης να επισημαίνουμε τις προσπάθειες τους για μείωση των δαπανών. Επαναλαμβάνω, όμως αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα, για την κυρία Χούμπνερ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Αν οι προτάσεις αυτές εφαρμοζόντουσαν μόνο σε επίπεδο ένωσης, θα είχαμε αύξηση της δραστηριότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε μείωση της ανταγωνιστικότητάς μας έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Το θέμα, η, η θέση αυτή είναι πολύ σύνθετη για μερικες κράτες κρά, κράτη-μέλη και θα το δείτε αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα μέτρα και αυτά τα εργαλεία, το FTT και το FAT, θα τα μπλοκάρουν. Από πληροφορίες που έχω σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. δεν θα υποστηρίξουμε μάλλον τροπολογίες που θέλουν επιπλέον φορολογικά έσοδα. Μεταφορά τους σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία δεν είναι απολύτως υπόλογα. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο ως κίνηση. Δεν συμφωνούμε με οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω δανεισμού από κράτη-μέλη και κυρίως από τους πολίτες τους, διότι ουσιαστικά οι πολίτες είναι οι φορολογούμενοι. Και στην έκθεση της κυρίας Ποδηματά φαίνεται ότι υπάρχουν υποδείξεις για αυτού του είδους το δανεισμό. Συμφωνούμε με το κείμενο που τονίζει την ανάγκη αναδιάρθρωσης των φορολογικών δημοσιονομικών πολιτικών και την εξηγίαση των εθνικών προϋπολογισμών επίσης και τον εξυγχρονισμό τους. Σας διαβεβαιώνω ότι η θέση μας έχει στόχο να αποφύγουμε την κοινωνική αναταραχή λόγω αναβολής εφαρμογής θεμελιωδών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε κάθε χώρα μέλος. Ευρωομόλογα. Μπορεί κάποιος να τα δει αυτά από διαφορετική ιδεολογική σκοπιά κάθε φορά. Και έτσι μπορεί να δει κανείς θετικά και να δει και αρνητικά σημεία. Δυσπιστώ όμως ως προς το ότι μπορεί τα ευρωομόλογα μειώνοντας τον ηθικό κίνδυνο να δώσουν μια λύση. Ίσως είναι ένας κρυφός τρόπος τα εθνικά χρέη να γίνουν ομοσπονδιακά, ας το πω έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος την αποτελεσματικότητα όλων των εργαλείων που ήδη έχουμε και το υπογραμμίζω αυτό, αντί να ψάχνουμε νέους τρόπους και πηγές. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας, κύριε Αποδηματά. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριο Κλούτε, θα λάβει το λόγο τώρα, αλλά θέλω να πω στην Κομισιόν ότι ο κύριος Επίτροπος μας είχε υποσχεθεί αυτή την έκθεση αντικτύπου όταν έγινε η ακρόασή του. Και τώρα μας λέτε το καλοκαίρι που έρχεται. Μου φαίνεται ότι έχει παρατραβήξει χρονικά αυτό για ένα απλό έγγραφο, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη γνώμη για τα θέματα αυτά. Κύριε Κλούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ποδηματά. Είναι πολύ καλή η δουλειά που έχει κάνει η σύνοψη πιθανών εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, κατά βάση αυτά τα οποία λέει η κυρία Ποδηματά είναι απαιτήσει της αριστεράς, ευρωομόλογα, φόρος διοξιδίου του άνθρακα, φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Βεβαίως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όπως λέμε. Η δεν συμβιβασμοί και ζητώ συγγνώμη, δεν είχα την ευκαιρία. Ε, είμαστε μικρή ομάδα, δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε όλες τις προθεσμίες, οπότε θα πρέπει να τις ξαναδούμε και να δούμε στις λεπτομέρειες τι μπορούμε να δεχτούμε. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ακόμη μια φορά το θέμα διεθνής ή πανευρωπαϊκός φόρος συναλλαγών Έχω καταθέσει και εγώ ίδιος μια τροπολογία πως θα ήταν λογικό να έχουμε ένα φόρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα απ' όλα για πρακτικούς λόγους κατά την άποψή μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δομές έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να εισαχθεί κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά μεγάλος οικονομικός χώρος οπότε μπορεί χωρίς μεγάλους κινδύνους να κάνει κάτι τέτοιο. Σε διεθνές επίπεδο είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Λείπουν οι ανάλογες δομές που θα μπορούσαν να μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο αποτελεσματικά και βραχυπρόθεσμα για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο για το πώς θα οργανωθεί είναι δύσκολο. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο είναι ευκταίο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Οπότε εμείς θα προτιμούσαμε, εάν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, να ξεκινήσουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κάτι το εφικτό, είναι ένας χώρος τον οποίο επηρεάζουμε άμεσα και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Κατόπιν να υποστηρίξω αυτό το οποίο είπε μόλις ο Φιλίπ Λαμπέρ. Δεν θέλω να το επαναλάβω. Απλά συμφωνώ και θα ήθελα να συμπληρώσω μία πτυχή. Ο Φιλίπ Λαμπέρ αναφέρθηκε στην πτυχή των επενδύσεων της στρατηγικής 2020. Να υπενθυμίσω, το είπα και χτες, πως πέρσι το έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού η Κομισιόν έχει υποβάλει μία πλατφόρμα και έχει ονομάσει εκεί πέρα, κατονομάσει πολύ φιλόδοξους ε, και αξιέπαινους στόχους και για να επιτευχθούν λοιπόν αυτοί οι στόχοι όπως αναγράφονται εκεί πέρα χρειαζόμαστε κονδύλια. Δεν γίνεται μόνο με οικονομία, δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για εξοικονόμηση και είναι αναγκαίο νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο για να διασφαλιστεί να αυτά τα κονδύλια ε, μακροπρόθεσμα για να ξέρουν και οι πολίτες ποια είναι η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ε, από αυτή τη σκοπιά θα έλεγα πως είναι αναγκαίο να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση οικονομική και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο στο επίπεδο των κρατών μελών. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Έχουμε 7 ακόμα λεπτά και έχω πέντε που θέλουν να αναλάβω το λόγο. Σας παρακαλώ να διαχειριστείτε με λιτότητα τον χρόνο σας για να μην καθυστερήσουμε. Η Βίκη Φόρντ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ στα project bonds, στα ευρωμόλογα για συγκεκριμένα σχέδια. Λέτε ότι οι τροπολογίες καλύπτονται στις συμβαστικές λύσεις. Αλλά εγώ δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνονται οι δικέ μου τροπολογίε απόλυτα στι συμβαστικέ τροπολογίε. Για μένα συμβαστική τροπολογία σημαίνει ή καλύπτεται τι τροπολογίε με λέξει κλειδιά όπω είναι οι δικέ μου τροπολογίε, ή αλλιώ πρέπει να ψηφιστούν χωριστά. Οι τροπολογίε μα λένε κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αμφιλεγόμενο για τα project bonds. Δεν λέει ότι είμαστε εναντίον των project bonds. Απλώς θεσπίζουν ορισμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ομόλογα. Η πρώτη τροπολογία, και αυτό έχει να κάνει και με τη συζήτηση που είχαμε κάνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πρώτο θέμα είναι το εξή. Αν έχετε σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, υπάρχουν ενδεχόμενες, ενδεχόμενοι κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να περάσουν από τη σωστή διαχείριση και τη σωστή δημοκρατική λογοδοσία. Θα μπορούσαν να τεθούν αυτά, τα, αυτή η διατύπωση στην συμβαστική τροπολογία. Αλλιώ πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά. Ένα δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα του αν υπάρχει ένα διαμεθοριακό ε, και διεθνικό σχέδιο να αντιμετωπίσουμε το θέμα του ηθικού κινδύνου. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη είναι πολύ ευαίσθητα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κοινέ εγγύησεις, δηλαδή οι φορολογούμενοι ενός κράτους εγγυούνται και για το άλλο κράτος, για το τμήμα του σχεδίου που είναι στο άλλο κράτος. Αν θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την ε, χρηματοδότηση με ευφυά τρόπο για, και να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του ενδεχομένου ηθικού κινδύνου, θα βελτιώσουμε την δυνατότητα. Και πάλι σας ζητώ ή να συμπεριλάβετε αυτή τη διατύπωση ή να ψηφίσουμε χωριστά. Και έτσι κι αλλιώς εγώ ε, ανησύχησα λιγάκι όταν αναφέρει ο Επίτροπος τα project bonds ως ε, financial engineering στα αγγλικά, δηλαδή ουσιαστικά χρηματοοικονομική μηχανική. Αυτό είναι μια έκφραση που δεν είναι ιδιαίτερα καλόδεκτη στη δική μου γλώσσα, το financial engineering. Επίσης ζήτησα ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπόκειται στα ίδια είδη διαφάνειας που θέλουμε, να υπάρχει επομένως και μια διαδικασία προβλέψεων κτλ. Εσεί, λοιπόν που υποστήριζετε πιο πολύ τη φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν γινόταν κάτι τέτοιο, να υπήρχαν προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, να, θα άλλαζε και, την, ε, και τη μορφή του προϋπολογισμού και ελπίζω να με υποστηρίξετε στι δικές μου τροπολογίε για μεγαλύτερη διαφάνεια στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αν συμφωνείτε. Ο κύριος Ούλμαν. Μπούλμαν μάλλον, συγγνώμη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Άννη Ποδηματά για το έργο που έχει φέρει σε πέρας, αλλά επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές, γιατί ξέρω πόσο επίμαχα είναι ορισμένα από τα σημεία αυτά και πόσο δύσκολο είναι να καταλήξουμε σε μια λύση των θεμάτων που είναι ακόμα ανοιχτά. Θέλω να σας υπενθυμίσω ποια είναι η βάση αυτής της συζήτησης και ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θέλουν να συζητήσουμε τα θέματα νέων πόρων, αλλά κύριε Φέρμπα θα σας ε, εκπλήξω ίσως λέγοντας ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία λοιπόν για την ε, επίσημη χρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έτος 2007, τότε θα καταλάβετε Αγαπητοί συνάδελφοι, και η κυρία Χιούμπνερ το γνωρίζει ήδη ως ε, εμπειρογνώμων στα θέματα αυτά, ότι είχαμε ήδη προχωρήσει σημαντικά στο επίπεδο αυτό Ήμασταν τότε σε ένα επίπεδο 60% υπερχρέωσης, τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο 80%. Επομένως, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταφέρει μεταξύ του 25 με 30% του ΑΕΠ τους, του συνολικού τους, ώστε να διασώσουν τράπεζες οι οποίες βρισκόταν σε μεγάλη δυσκολία. Ξαναλέω, 25 με 30% του ΑΕΠ. Αυτό σήμαινε και μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και πτώση του συνολικού ΑΕΠ σε, σε επίπεδο 4 και 5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μας έχει φέρει στην κατάσταση αυτή λόγω της ισόρευσης του χρέους. Μπορεί κανείς να ψάξει τώρα τους υπευθύνου όπου θέλει, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι δραματικού χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας πει ο κύριος εκπρόσωπος της Κομισιόν αυτά που έλεγε ο Επίτροπος Σέμετα. Η κατάσταση είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία δεν αντιμετωπίζεται με τα μέτρα αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Και θέλω να πω, κυρία Χιούμπνερ, αν το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή ακολουθήσει την αδράνεια της Κομισιόν και του Συμβουλίου, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι δεν θέλω να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά αν ακολουθήσουμε μια τέτοια αντιμετώπιση, μετά από μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει καμία συνοχή μέσα στην ευρωπαϊκή ζώνη. Θα είναι μια τελείως διαφορετική ζώνη πλέον. Θα μπορούν να μπουν άλλες χώρες, αλλά κάτω από διαφορετικές συνθήκες ίσως. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε αποφασιστικά μέτρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να μπορέσει να επομιστεί τις ευθύνες που έχει έναντι των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν ότι η θέση που ανέφερε σήμερα το ΕΛΚ δεν είναι η τελική του λέξη. Ευχαριστώ τον κύριο Σμιτ για την ευκαμψία που έχει δείξει στο θέμα αυτό και ελπίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αν είναι λοιπόν η τελική σας στάση του ΕΛΚ, μήπως θα έπρεπε να επανέλθουμε στην ανάγκη που ε, υπογραμμίζει και η κυρία Βόρτμαν Κόλ, η Κομισιόν επιτέλους να δώσει αυτή την έκθεση αντικτύπου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην απαραίτητη νομοθεσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούμε να είμαστε εκτός χρονικού ορίου. Το πρόσφορο είναι και σύντομο, όπως λέμε στα, στα ισπανικά. Ο κύριος Φέμπερ. Ευχαριστώ. Σωστά αναφέρατε ήδη πως ε, μας είχε υποσχεθεί ο Επίτροπος μία ε, μελέτη επιπτώσεων ήδη πριν από ένα έτος ε, πέρσι τον Φεβρουάριο στην Ολομέλη. Οπότε κύριε Μπούλμαν, αν μιλάτε για καθαίριση μην απευθύνεστε σε εμά, απευθυνθείτε στην Κομισιόν. Δεύτερον, το θέμα το οποίο συζητάμε αναφέρεται καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και δεν ξέρω εάν οι νέοι φόροι είναι τίποτα το καινοτόμο. Και βεβαίως κύριε Λάμπερτς μία απάντηση ξέρετε μόνο ε, αυτή των ε, πρασίνων αλλά βεβαίως εμείς έχουμε άλλη απάντηση και ευτυχώς γιατί αλλιώς ήταν βαρετά τα πράγματα. Κοιτάξτε η απάντηση είναι απλή αν ισχύουν αυτά τα οποία λέτε θα πρέπει να παραδεχτείτε πως πρέπει να ανατρέξουμε όλο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τον... Ε, η απάντηση δεν είναι επειδή είναι χρεωμένα τα κράτη να χρεώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωομόλογα. Η απάντηση είναι πως ε, εάν ε, δεν μπορεί πλέον, πλέον η Ελλάδα να πληρώσει ένα ποσοστό 10% σε επιτόκια όπως πλήρωνε επί ε, και πληρώνει 3,5% πρόκειται για μια τεράστια εξοικονόμηση. Αυτό είναι το θέμα και μην λέμε πάνε τα πράγματα στραβά και πρέπει να μοιραστούν το βάρος οι υπόλοιποι. Δεύτερον, τα προβλήματα των υπερχρεωμένων προϋπολογισμών ε, δεν λύνονται με το να αρχίσουμε να συσσωρεύουμε άλλα χρέη σε άλλο επίπεδο. Πρέπει να απαντήσουμε τελείως ήρεμα το θέμα τι είναι η αποστολή του κράτους στον 21ο αιώνα και εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι ένα κράτος ε, το οποίο θα παρέχει τα πάντα, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα λεφτά. Εάν βεβαίως είναι το κράτος το οποίο πιστεύει στην ατομική ευθύνη, υποστηρίζει την ε, οικονομική δραστηριότητα, τότε χρειαζόμαστε λιγότερα λεφτά. Η απάντηση λοιπόν δεν μπορεί να είναι προχωράμε προς τα μπρος και επιβάλλουμε νέους φόρους και ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα καλά. Θα είμαι σύντομη λόγω του, του χρόνου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον Ανυποδηματά και τους σκιώδησηγητές για την προθυμία τους, γιατί είναι προφανές πως έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Την θέλησή τους λοιπόν να βρουν συμβαστικές λύσεις και οπωσδήποτε το αποτέλεσμα που θα ήθελα εγώ να δω είναι να έχουμε Ανοιχτέ απόψεις στο Σκηνοβούλιο για καινοτόμους τρόπους ε, φορολόγηση και εσόδων. Γιατί, γιατί αλλάζουν ε, τα πράγματα στον, στον κόσμο και δεν είναι λογικό από εμάς να έχουμε μία παραλυμένη, απολυθωμένη άποψη και να λέμε δεν το θέλουμε. Να Πόσους συναδέλφους από την δεξιά. Αν σας αποδεικνύαμε πως δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στα κέρδη, θα λέγατε ναι, γιατί αυτός είναι ο μόνος όρος που έχετε. Ε, γι' αυτό δεν το θέλετε. Και μάλιστα κάποιες έρευνες λένε πως σε ένα απειροελάχιστο επίπεδο δεν θα έχει αντίκτυπο ε, στα κέρδη και στα μπόνους που θα πληρώσουν ε, οι τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποφάσισε η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα. Δεν θα υποφέρει ο τραπεζικός τομέας γιατί θα φροντίσουν για την ανταγωνιστικότητά του ακράτη μελη Να σας υπενθυμίσω επίσης συνάδελφοι πως και εγώ αναμένω, σε... αναμένα κάρμουνα την αξιολόγηση της Κομισιόν αλλά δεν περιμένω και πάρα πολλά γιατί ήδη η Κομισιόν έχει αποκλείσει τέτοιο φόρο χωρίς να κοιτάξει καν τα στοιχεία. Είπε όμως πως ω κλάδος οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν φορολογείται αρκετά σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Έχει λάβει 3 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, όχι μικροποσά, και αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς, η δική μας πλευρά, είναι πως θέμε και λίγη δικαιοσύνη. Πρέπει να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί, να στηρίξουν την οικονομία και ελπίζω το αποτέλεσμα αυτού του συμβιβασμού να είναι να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα όπως κάναμε και με την έκθεση Μπερές, πως πρέπει να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί. Όχι να του πάρουμε τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά του, δεν σημαίνει αυτό. Πρέπει να συνεισφέρουν στην πραγματική οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και αν καταλήξουμε σε τέτοιο συμβασμό, οπωσδήποτε θα υπερψηφίσω. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ. Ζαν Πολ. Κύριε Πρόεδρε, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που στόχο θα πρέπει να έχουμε όχι να κάνουμε μια έκθεση ακόμα να την βάλουμε σε ένα ράφι να σκονίζεται, αλλά να κάνουμε μια έκθεση όπου το Κοινοβούλιο να τονίζει τις θέσεις του. Νομίζω η δεύτερη λύση είναι πιο σωστή και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Πρόεδρος, πολύ σωστό αυτό που είπατε. Ηλικό. Πράγματι είναι δύσκολη κατάσταση και μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, αλλά δεν υπάρχουν εδώ πέρα οι βάσεις για την ε, λήψη απόφασης. Είχε έρθει χτες εδώ πέρα ο Ούγγρος υπουργό και ήταν επιφυλακτικός εκεί που θα μπορούσε να έχει απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί είναι απλό. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ναι. Πράγματι βλέπετε πως ε, κινδυνεύει η πραγματική οικονομία από την αύξηση των ε, συναλλαγών αυτών των χρηματοοικονομικών. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία στο πλαίσιο των G20 δεν σημαίνει πως είναι κάτι το καινοτόμο η φορολογία αυτή. Η καινοτομία δεν είναι πάντα άλλος ένας φόρος. Αντιλαμβάνομαι πως βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις γρήγορα και η πρόεδρος ανέφερε χτες πόσο γρήγορα πρέπει να αποφασίσουμε. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε το ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση δεν θα έχουμε ε, λάθος αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσει η Κομισιόν να υποβάλει γρήγορα τη σχετική της μελέτη. Μετά βεβαίως έχουμε και την ε, τροπολογία 24 στην παράγραφο H όπου λέμε πως ε, το σύμφωνο σταθερότητας ε, είναι ένα μέσο και όχι ένας ε, αυτός Και βεβαίω ε, το θέμα της λειτουργίας του σχετίζεται με τους ελέγχους και το τι έγινε σε κάποιες χώρες. Τι πρέπει λοιπόν να πούμε τα πράγματα χήμα, να ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι για αυτή την κρίση για να κινηθούμε και ανάλογα προς το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω άλλου δύο οι οποίοι θέλουν να ζητήσουν το λόγο. Ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι επειδή θέλουν να κάνουν μια ε, παρατήρηση επί προσωπικών θεμάτων. Ο κύριο Λάμπερτ, ο οποίο είναι γνωστό για την ευγλωτία του, καταρχήν βεβαίω. Σε 30 δευτερόλεπτα να απαντήσω στον Μάρκο Φέρμπερ. Είσαι πολύ, ήσουν πολύ σαφή ότι ουσιαστικά ο στόχο σα είναι να μειωθεί το κράτος και να δοθεί περισσότερο χώρο στον οικονομικό στίβο στι επιχειρήσει, Αλλά βλέποντα τη δική σα χώρα, η οποία είναι ο καλύτερο μαθητή στην Ευρώπη, αυτό που μα οδηγεί. μα οδηγεί σε ένα ιδιογκωμένο χρηματοοικονομικό χώρο και 7 εκατομμύρια Γερμανοί εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι σε επισφαλείς συνθήκες. Το ερώτημα το οποίο μπορούσαμε να μου στο διάδρομο Πού νομίζω θα βρει πελάτες η επιχείρηση, το επιχειρήν στη χώρα σου, αν ο κόσμος γίνεται τόσο πιο πολύ, πιο φτωχότερος. Λοιπόν, στην ώρα του καφέ θα συζητηθεί αυτό το πράγμα. Ο κύριος Σμιτ. Η κόρα μου δεν, δεν πηγαίνει άσχημα σε αυτό το παιχνίδι. Ε, και δεν έχουμε τόσους φτωχού εργαζόμενους. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ε, απεσιόδοξος για τα θέματα αυτά θα κάνει προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Ζώνη για να τα λύσει αυτά τα θέματα και μετά χώρες όπως η Πολωνία και η Σουηδία μπορεί να έχουν προβλήματα να είναι εκτός της Ευρωζώνης και να θέλουν να μπουν. Είμαι πιο αισιόδοξο λοιπόν από τον κύριο Μπούλμαν για τα θέματα αυτά, γιατί η εναλλακτική λίστα είναι ολέθρια. Εγώ είμαι υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας και των θεμάτων αυτών αλλά δεν είμαι πεπισμένο για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και για την κυρία Χίμπνερ θα ήθελα να πω ότι εμείς υπερψηφίσαμε τελικά την έκθεση Μπέρες, αλλά κρατήσαμε μια διαφοροποιημένη θέση σε σχέση με το θέμα της επιβολής του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών μόνο στην Ευρώπη. Γι' αυτό ίσως μπορούμε να παραμείνουμε και σε αυτή την έκθεση σε αυτό το επίπεδο. Προτού πίσω τους άλλους εξοργισμένους συναδέλφους στην ομάδα μου θα θέλω να ξέρω αν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Τι τυχερός που είσαστε κύριε Σμιτ. Λοιπόν, τελειώνει αυτό το το διάστημα συζήτησης. Ναι, Ντανούτα, σύντομα παρακαλώ. Μα αν αναφέρετε το όνομά μου το οποίο μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα, θέλω να απαντήσω σε αυτά τα θέματα. Ξεχνάμε ότι σε αυτή την έκθεση τη κυρία Ποδηματά δεν συζητάμε να το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αλλά και άλλε διαδικασίε, άλλε μορφέ φορολογίε, παραδείγματο χάρη ενεργειακού φόρου κτλ. Πρέπει να πω ότι πολλέ φορέ είμαστε προσδεδεμένοι σε διαφορετικέ οικονομικέ θεωρίε ο καθένα μα. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ότι χρειάζεται για την ανάπτυξη στην Ευρώπη που είναι η κύρια μέρημνά μα ότι χρειαζόμαστε σημαντική χρηματοδότηση και αυτή η χρηματοδότηση θα έρθει και από το δημόσιο τομέα. Όπω είναι οι εθνικοί προπολογισμοί και ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Και λέω ότι λόγω των περικοπών στο δημόσιο τομέα και τη κατάσταση η οποία επικρατεί <clears throat> και βλέπουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο προδιαγράφεται ότι αυτά τα οποία θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα που είναι κυρίως ο τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας θα παίξουν ένα προεξάρχοντα ρόλο. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου εξάλλου ότι όταν σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε εργαλεία δημόσιας πολιτικής αυτά τα εργαλεία στο ελάχιστο δεν πρέπει να υπονομεύουν και να υποσκάπτουν τη δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να δώσει την κατάλληλη χρηματοδότηση η οποία θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. <clears throat> και επίση πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σχεδόν πεπισμένοι ότι αν εφαρμόσουμε νέα καινοτόμα εργαλεία αυτό θα οδηγήσει σε καθαρή αύξηση τη δυνατότητα επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων. Αν δούμε τι γίνεται τώρα στις κεφαλαίες αν δούμε πού πηγαίνουν τα κεφάλαια, αν δούμε τον τραπεζικό τομέα, και εγώ βλέπω με μεγάλη ανησυχία τις, ε, τα στρες τεστ των τραπεζικό τομέα και τα θέματα της ρευστότητας. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για ανάπτυξη με το να εφαρμόσουμε φόρους όπως ο φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Γι' αυτό δεν είμαι πεπισμένη και γι' αυτό πολλοί από τους συναδέλφους του ΕΛΚ εξακολουθούν να είμαι πεπισμένοι. Γι' αυτό εμείς προ προτάσουμε την ιδέα του να περιμένουμε τέσσερις μήνες ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε από την Κομισιόν μια σαφή απάντηση. Μπορεί να είναι λαθασμένη αυτή η απάντηση, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε μια βάση επί της οποίας να στηρίξουμε την απόφασή μας, να έχουμε κάποιο σημείο αναφοράς και δεν θα έχουμε απλώς πολιτικά μηνύματα, κάτι το οποίο κατανοώ ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από τις πολιτικές μας απόψεις για αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σίλβι Γκουλάρ, θα σου δώσω το λόγο, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Και έχουμε και άλλα σημεία στη μέση διαταξή. Καταρχήν είναι θετικό το ότι πολλοί συνάδελφοι προσπαθούν να πετύχουν μια σύγκληση. Κάτι όμως που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι όταν λέμε ναι συμφωνούμε συνολικά ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πετύχουμε ένα μέτρο σε τέτοιο επίπεδο. Μην ξεγελάμε τους εκλογείς και τους πολίτες. Αν λέμε ναι γίνεται με υπέρ σε γενικό επίπεδο που λέμε στα Ισπανικά μανιάνα μανιάνα. Αύριο θα γίνει, αύριο θα γίνει, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Α δεχτούμε ότι, να πούμε ναι ότι οι αγορέ συνολικά έχουν μια επίπτωση στην πολιτική μας ημερήσια διάταξη. Περί αυτού πρόκειται. Και όχι ότι τα κράτη-μέλη και η Ένωση μπορούν να ξεπεραστούν από την τεχνολογία, από τι εξελίξει. Τι θέλω να πω. Προσωπικά προτιμώ να μείνουμε στο ότι έχουμε ένα αλφα περιθώριο ελιγμών και το δεύτερο που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το ζητάμε ένα σωρό εκθέσεις από την Κομισιόν. Και μετά τι γίνεται με τις εκθέσεις αυτές. Την περασμένη εβδομάδα συζήτηση για τον ανταγωνισμό. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά πάνε σαν άνθρωπο που μου. Ο Επίτροπος Αλμούνια δεν ήρθε. Ζητήσαμε ήδη και πέρυσι διάφορα πράγματα. Καμιά απάντηση. Μην γίνουμε εδώ ένα κλαμπ, ένα όμιλο ανθρώπων που ζητάμε από εκθέσει από την Κομισιόν και η Κομισιόν με τίποτα αδιαφορεί τελείω. Μα γράφει τα παλιά τη τα παπούτσια. Πολύ ενδιαφέρον σε έκθεση συναδέλφου κυρία Ποδηματά. Η καινοτομία μπορεί να έγκυται, να στηριζόμαστε, να βλέπουμε τα λεπτά σημεία του τι χρειάζεται. Όταν πάρουμε όμω το Annual Growth Survey και δούμε την πρόταση τη Κομισιόν που λέει μόνο να αυξηθεί ο ΦΠΑ, τότε τι να πω. Ξεχάσαμε την έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης. Πρόεδρος, θα στείλει κάποια επιστολή η Κομισιόν για το θέμα αυτό. Μάλλον εμείς θα στείλουμε μια επιστολή στην Κομισιόν ως Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων λέγοντας ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της απάντησης στα ερωτήματά μας. Ή αν έχει και πάλι το λόγο. Για δύο λεπτά μόνο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλους ε, για, τις, ε, για τη συμβολή τους, για τα όσα είπαν. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, ότι ε, πιστεύω και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα είναι και περιεκτική και που θα υπερασπίζεται τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα αυτού του σώματος. Δύο λόγια μόνο, συμπυκνώντας τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν σε σχέση, με τα, ε, σε σχέση με τα ευρωομόλογα, τα ευρωομόλογα όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά δεν είναι μια καινούργια ιστορία ούτε είναι μια ιστορία που επινοήθηκε τώρα στο πλαίσιο της κρίσης χρέους από κάποια υπερχρεωμένα κράτη προκειμένου να μεταθέσουν το βάρος του το, του χρέους τους κάπου αλλού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά, ε, για μια ιδέα που ε, χρονικά συμβαδίζει με την γέννηση και τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θυμίζω ότι, ότι προπομπός αυτής της ιδέας αποτυπώνεται στο, στην έκθεση Τζοβανίνη του Νοεμβρίου του 2000 όπου θεωρείται τότε ε, η έκδοση ευρωομολόγων ως σημαντικό εργαλείο για την ολοκλήρωση της αγοράς ε, και για την ενίσχυση της Ένωσης δεν προχώρησε για λόγους πολιτικού συσχετισμού στο Συμβούλιο. Επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο. Προφανώς οι λόγοι για τους οποίους επανέρχεται έχουν να κάνουν και με την ε, εκτεταμένη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ε, ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Νομίζω ότι ε, αξίζει τον κόπο συνυπολογίζοντας προφανώς όλες τις παραμέτρους να εξετάσουμε σε βάθος αυτήν τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, όχι για να μεταθέσουμε το βάρος της ευθύνης από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό, από τους αδύναμους στους ισχυρούς, αλλά για να δώσουμε μια δυνατότητα στην Ένωση να βγει το συντομότερο δυνατό από την κρίση και να διευκολύνουμε και να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται ε, στο εθνικό επίπεδο από μια σειρά χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξηγειάνουν τα δημόσια ε, οικονομικά τους. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και η διαπραγμάτευση για την οικονομική διακυβέρνηση, μια σειρά ποινές και κυρώσεις που συζητάμε σήμερα, εκτός από τις ποινές και τις κυρώσεις, επειδή δεν απευθυνόμαστε μόνο σε κυβερνήσεις, απευθυνόμαστε και σε πολίτες, διότι οι πολίτες είναι αυτοί που αναλαμβάνουν σε τελευταία ανάλυση το βάρος της εφαρμογής όποιων πολιτικών επιλογών. Οι πολίτες, για να μην ε, ε, απομακρυνθούν από την ευρωπαϊκή ιδέα, είτε προέρχονται από κράτη-μέλη με προβλήματα, είτε προέρχονται από κράτη-μέλη ε, δυνατά, ε, με υγιείς οικονομίες, ε, έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους σήματα. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να ξανανοίξω την κουβέντα σε σχέση με το, την υπόθεση του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο ευρωπαϊκό ή στο παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει νόημα. Άλλωστε, ούτε η έκθεση αυτή ε, έχει την πρόθεση να δώσει απάντηση στο τεχνικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχουν διάφορες παράμετροι, διάφορες τεχνικές πτυχές. Η δουλειά μας και ο ρόλος μας όμως εδώ είναι πολιτικός καταρχήν. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και που πρέπει να πετύχουμε κατά τη γνώμη μου είναι να δώσουμε ένα ισχυρό πολιτικό σήμα ότι θα πρέπει ε, αυτή η, η προοπτική, αυτή η δυνατότητα να διερευνηθεί γρήγορα και στα σοβαρά είναι προφανέ ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρώπη εάν δεν έχει προηγηθεί μια μελέτη επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι εκ των όνου κάνευ. Πολιτικά όμω εμεί πρέπει να δώσουμε ένα σήμα. Σήμερα ακόμα περισσότερο, διότι η Γαλλία έχει αναλάβει την προεδρία του G20, η Γαλλία έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν υπέρ ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, Λοιπόν, είναι, νομίζω, επιβάλλεται από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά του Κοινοβουλίου και της Ένωσης συνολικά, αποδεικνύοντας ότι είναι συνεπής προς τις θέσεις που έχει πάρει κατά καιρού. Ε, να ε, επαναλάβουμε ε, ότι θα πρέπει να προχωρήσει να γίνουν σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και προκειμένου να ασκηθεί με αποτελεσματικό τρόπο πίεση στο παγκόσμιο επίπεδο η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα όπως το έχει κάνει στο παρελθόν. Πολιτικά ξαναλέω, το τεχνικό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ελπίζω ε, να καταφέρουμε να καταλήξουμε κάπου τις ε, ημέρες που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ε, Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου για να είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ξέρω ότι είναι σαφή η θέση των πολιτικών ομάδων, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επιμείνουμε στο να διατυπωθούν αυτές τις θέσεις, αλλά απλώ πρέπει να γίνει προσπάθεια εξέβρεση συμφωνίας εφόσον αυτό είναι εφικτό. Λοιπόν, κλείνω αυτό το σημείο της ημέρας διάταξης, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης, το οποίο είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2009 με εισηγητή τον κύριο Σαμπίν Κούτασο. Λυπάμαι κύριε Κούτα για την καθυστέρηση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος έτσι ώστε να τελειώσουμε εγκαίρως μέχρι τις 10.30. Η ετήσια έκθεση λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μια ανάλυση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας το 2009. Προτείνουμε κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές δράσεις της Τράπεζας. Είναι σημαντικός εταίρος της Ένωσης για τους πολιτικούς στόχους αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης που ζούμε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε για οικονομική σταθερότητα και οικονομική ανάκαμψη. Τονίζω την σημασία του ρόλου της τράπεζας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020 με έκδοση ειδικών ομολογιών και με σύνταξη προγραμμάτων που θα δημιουργήσουν απασχόληση συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων που έχουν στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποδομή ε, της ενέργειας και των μεταφορών. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, η τράπεζα απέκτησε ένα βαθμό ευελιξίας για τις διάφορες μορφές δράσης της. Η τράπεζα από εδώ και μπρος της επιτρέπεται να προσφέρει τεχνική βοήθεια, να δημιουργήσει θυγατρικές μονάδες, τεχνική βοήθεια κυρίως σε τομείς στόχων σύγκλησης. Θα ακούσω με πάλι πάρα πολύ προσοχή τη γνώμη των συναδέλφων. Όσον αφορά δε το χρονοδιάγραμμα, προθεσμία για τροπολογίας 7 Φεβρουαρίου, συζήτηση των τροπολογιών στην Επιτροπή μας στις 28 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία 15 Μαρτίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια 4 Απριλίου. Ευχαριστώ. Κυρία Χούμπνερ και εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Δεν νομίζω ότι όπως λέγανε ορισμένοι ότι αυτό είναι ένα θέμα ρουτίνας business as usual. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω της χρονικής στιγμής στην οποία έρχεται. Έρχεται σε μια ε, χρονική στιγμή όπου έχουμε τα προβλήματα με τα σχέδια λιτότητος, με την πολυετή δημοσιονομική σχεδίαση και την αναζήτηση πηγών οικονομικής ανάπτυξης. Από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να δούμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα στη μελλοντική εμπλοκή της ΕΤΕ στο να διευκολύνει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, την ε, μόχλευση ουσιαστικά που προέρχεται από τη χρήση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει ανάπτυξη και χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης το γεγονός ότι η ΕΤΕ έχει κάνει σημαντική συνεισφορά στην απάντηση της, κρίσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της κρίσης ακριβώς με το να επιτρέψει να υπάρχει μια χρηματοδότηση με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Έχουν γίνει πολλές κοινέ χρηματοδοτικές προσπάθειες και εργαλεία μεταξύ Κομισιών και ΕΤΕ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη δυνατότητα αυτή πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων χάρη στη συμμετοχή της Κομισιόν και της ΕΤΕ και το ψήφισμα αυτό τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΤΕ για την διευκόλυνση της χρήσης του προϋπορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των επενδύσεων στα επερχόμενα χρόνια. Για όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε σε αυτό το ψήφισμα τις επιτυχίες οι οποίες έχουν προέλθει <clears throat> από τη δράση της ΕΤΕ και την επιτυχία της ΕΤΕΣΤΟ να προχωρήσει σε πιο ε, σημαντικές μορφές χρηματοδότηση, ιδίω στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής, την υποστήριξη των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αστικών, ε, της ανανέωσης του αστικού χώρου, πρωτοβουλίες όπως Jasmine, Jessica κτλ. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό Ιδιαίτερα επέκεινα το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν και να πολλαπλασιάσουν αυτές τις πρωτοβουλίες, ιδίως συνδυάζοντας τις χορηγήσεις από τις ευρωπαϊκές πολιτικές με χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή τις ε, χρηματαγορές εν γέννη. Και στο πλαίσιο αυτό Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τη σημασία των λεγόμενων project bonds, λαμβάνοντα υπόψη αυτά που είπε προηγουμένως η Βίκη Φόρτ για τα θέματα διαφάνειας. <clears throat> Πιστεύω ότι τα project bonds, τα ευρωμόλογα για συγκεκριμένα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνονται ότι είναι ένας από τους καλύτερους δρόμους προς τα εμπρός για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες επενδύσεων υποδομών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν υπολογίζει ότι θα χρειαστούμε περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ για τις υποδομές μεταφορών. Αυτά δεν μπορούν να βγουν από κρατικούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να υποστηριχθούν <clears throat> μέσω project bonds από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και εγώ θα καταθέσω λοιπόν μία ή δύο τροπολογίε με στόχο να ενισχύσουμε το, το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υπάρξει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε το ρόλο τη ε, ΕΤΕ στο να δημιουργήσει τα εργαλεία αυτά τα οποία θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις για ε, υποδομές στις ε, τηλεπικοινωνίες και στη μεταφορά και στον ενεργειακό τομέα που μέχρι στιγμή είχαν αντιμετωπιστεί μονάχα με άμεση <clears throat> χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, κάτι το οποίο στι τωρινέ συγκυρίε δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικό. Γι' αυτό θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτό το ψήφισμα στο τωρινό πλαίσιο. Κύριε θέλετε τον λόγο. Γιούργεν. Όχι, Έπινγκ δεν είναι εδώ. Ο Σβέν. πήγαν πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Κοιτάξτε, δεν σημαίνει αυτό όπως το πρόσωπο τους φιλελεύθερους, αν και έλαβα κάποια περίεργα email από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεση. Ένα γενικό σχόλιο. Θα ήθελα να ξανασκεφτούμε πώς μπορούμε να πλησιάσουμε το, το 2009 υπάρχει ένα θέμα διαδικασίας, δεν ξέρω, ίσως οι παλαιότεροι συνάδελφοι μπορούν να μου εξηγήσουν πώς εν έτη 2011 συζητάμε το 2009, κάτι το οποίο μου φαίνεται περίεργο δεδομένη της κρίσης. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας και θα ήθελα να τονίσω πως ειδικά το κομμάτι για τη χρήση ε, χρηματοδοτικών μέσων υπερακτίων και των φορολογικών παραδείσων με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και ελπίζω να μπορέσουμε να ενισχύσουμε έτσι τις εξελίξεις που λαμβάνουν ήδη χώρα στην Τράπεζα Επενδύσεων προς αυτό. Γενικότερα νομίζω πως αυτό το οποίο λείπει από την έκθεση και θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω να συνεργαστούμε είναι το εξής. Νομίζω ε, η περιβαλλοντική διάσταση των νέων επενδύσεων και οι στρατηγικές ανάπτυξης λείπουν. Βεβαίω αυτή είναι η παραδοσιακή ρόλη που έχουν οι πράσινοι ε, για το πρασίνισμα της οικονομίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Χρειάζονται κάποια κεφάλαια όταν μιλάτε για ομόλογα έργων στις παραγράφους 11 με 13 θεωρούν πως αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα για να έχουμε έναν οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας. Όταν μιλάμε για, για την παράγραφο 17 είναι πολύ γενική η παρατήρηση το να λέμε πως ε, όλα τα διευρωπαϊκά δίκτυα και η υποδομή των μεταφορών είναι κάτι του οποίου είμαστε υπέρ. Και πάλι πρέπει να αφορά ιδιαίτερα αηφόρες μεταφορές. Δεν έχει νόημα να επενδύουμε τεράστια ποσά σε υποδομές οι οποίες δεν συμβιβάζονται με τις ανάγκες κλιματικής αλλαγής. Σπαταλάμε λεφτά. Οπότε πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό εκεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρούμε σημαντικό είναι να ευθυγραμμίσουμε την συμπεριφορά της τράπεζας όταν μιλάμε για χρηματοδότηση της ενέργειας. Ευτυχώς τονίσατε πως θα πρέπει να δώσουμε βάρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά περιοριζόμαστε στις αναψώμενες χώρες. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να πάμε ε, σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως δεν συμβιβάζεται με κάποιες επενδυτικές συμπεριφορές της τράπεζας. Οπότε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρουσιάζει αυτόν ως υποστηρικτή των ανανεώσιμων, αλλά ταυτόχρονα χρηματοδοτεί έργα που πάνε αντίθετα με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης που έχουμε ψηφίσει το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι επένδυση της τράπεζας στο, σε λιγνητορυχείο στην ε, Σλοβενία, στο οποίο έδωσε 550 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν ελπίδες για φιλόδοξη κλιματική πολιτική στην Σλοβενία για να μειωθούν κατά 80% οι εκπομπές μέχρι το 2050 για να μειωθεί, για να παραμείνει η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Όλη η ποσόστοση εκπομπών της Σλοβενία θα συνεχιστεί με την λειτουργία αυτού του εργοστασίου, θα απορροφηθεί από αυτό το εργοστάσιο. Οπότε χρηματοδοτούμε εδώ πέρα κάτι αντίθετο με αυτό το οποίο ψηφίσαμε εδώ πέρα και έχουμε δεσμευτεί ε, διεθνώς για την κλιματική πολιτική. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή επενδυτική συμπεριφορά. Πέρα από αυτό, Νομίζω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως θέλουμε σαφέστερες αναφορές ε, όσον αφορά το πώς χρησιμοποιούνται τα λεφτά, δηλαδή να πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο σε μεγάλες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Επιπλέον θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς ε, θα βελτιωθούν οι μεσοπρόθεσμες αναφορές και Τέλο πάντων, για να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο, αυτά είναι κάποια από τα βασικά ζητήματα για εμά. Αηφορία και σαφής ευθυγράμμιση πρασίνων προδιαγραφών και προδιαγραφών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επενδύσεις τη Τράπεζα. Ναι, συγγνώμη, δεν είχα όλο τον κατάλογο των ε, σκιωδών, εξού και η περίεργη σειρά που ακολούθησε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ τον κύριο Κούτας για την εργασία του στο σχέδιο έκθεσης. Συμφωνώ και εγώ με την ανάγκη να ενισχυθεί το έργο της τράπεζας όσον αφορά τον δανεισμό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης συμφωνώ με τον εισηγητή να προσανατολιστεί με το πώς θα προσανατολιστεί η τράπεζα στο μέλλον για να έχουμε μεγαλύτερη μακροοικονομική σύγκληση μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Όπως ξέρετε πέρσι, πολλές χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης έχουν τα προβλήματα που γνωρίζουμε. Χώρες του Νότου αντίθετα έχουν τα προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με το πρόγραμμα της τράπεζας. Επίσης συμφωνούμε με την ανάγκη η τράπεζα να εκδίδει ομόλογα προκειμένου να ενισχύονται υποδομές ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Θα πρέπει να έχει προτεραιότητα στη χρήση μεθοδολογίας όπως η λεγόμενη ανάλυση κόστος ωφέλους προκειμένου στα συγκεκριμένα προγράμματα να έχουμε τον μεγαλύτερο πολυπλησιαστικό αποτέλεσμα σε όρους ΑΕΠ. Στα ενεργειακά προγράμματα που αναφέρει ο εισηγητής θα πρόσθετα και προγράμματα για την μεταφορά φορτίων με τρένα. Και πιο συγκεκριμένα, μια από τις προτεραιότητες της τράπεζας θα έπρεπε να είναι τα διασυνοριακά δίκτυα φορτίο που να φτάνουν στα μεσογειακά λιμάνια. Αυτό θα τα συνέδε έτσι με τις ευρωπαϊκές αγορές και θα βελτίωνε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τώρα για τον αναπτυξιακό ρόλο της τράπεζας. Αν και Χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Καλό θα είναι να γίνεται και καλύτερη συνεργασία με ε, προσωπικό επιτόπια έτσι ώστε η τράπεζα να ασκεί τον διοικητικό ρόλο σε συνεργασία και συμφωνώ με τους κύριους στόχους και τις πεσνές δραστηριότητες της τράπεζας ιδιαίτερα τώρα που ορισμένες χώρες στην Ένωση έχουν σοβαρά πιστοτικά προβλήματα. Ο Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για την έκθεση. Ως πρώην εισηγητής για την τράπεζα μπορώ να εκτιμήσω την καλή ποιότητα της δουλειάς του συναδέλφου. Αλλά η τράπεζα ΚΑΤΕΜΕ δεν είναι για να δρά προδραστικά Να πούμε δηλαδή ζούμε τη χειρότερη κρίση από τη δεκαετία του 30. Και αυτό θα έπρεπε να κάνει η τράπεζα αυτή. Θα έπρεπε να υπάρξει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρόεδρου Βανδρομπάη και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή κάτι τέτοιο ή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μερικές σύντομα σημειώματα από τον επικεφαλής της τράπεζας πέρα από, την, από τις επενδύσεις μακροοικονομικού χαρακτήρα που δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικές αλλά τι προστιθέμενη αξία έδωσαν στην κρίση που ζούμε. Ξέρουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρουμε τι κάνουν τα άλλα θεσμικά όργανα. Δεν ξέρουμε αρκετά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να προσφέρει πολύ πιο σοβαρό έργο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, ναι, να μελετήσουμε την έκθεση του 2009 για να δούμε τι έγινε, αλλά σε σχέση με τα δεδομένα τα τώρα και για το μέλλον χρειαζόμαστε περισσότερα μακροοικονομικά στοιχεία. Θα θέλαμε ο πρόεδρος της τράπεζας αυτής όχι να έρθει εδώ σε μια ακρόαση, ας μας στείλει μερικές σελίδες, σημειώματα, να μας πει τι κάνει σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, σε μακροοικονομικό επίπεδο, προκειμένου να φέρει σε πέρας σωστά το έργο της και να παίξει σωστά το ρόλο της. Δεδομένη της κρίσης στην οποία ζούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Έχουμε έναν εκπρόσωπο της τράπεζας εδώ τώρα, τον κύριο Κρένκορς. Δεν ξέρω αν θέλει να μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο, απάντηση. Αν θέλει, ένα λεπτό. Ένα λεπτό δίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για το εξαιρετό έργο του και την καλή συνεργασία που είχαμε. να τονίσω πρώτα απ' όλα που συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις κυρίας Χούμπνερ για τη σημασία των νέων ε, χρηματοοικονομικών μέσων. Θα χρησιμοποιούσα τρεις λέξεις ε, που επανέλαβε ο πρόεδρος, ο κύριος Μέιστατ, πως θα πρέπει να είναι απλά τα νέα μέσα, για να είναι διαφανή, να παίζουν καταλητικό ρόλο για να φέρνουν και άλλους φορείς γύρω από το τραπέζι και βεβαίως θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το χρήμα στο μέγιστο βαθμό. Οπότε για τον κύριο Κιγκό πράγματι παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα οποία είπε. Είχε έρθει στο Λουξεμβούργο πρόσφατα για να συζητήσουμε αυτά τα έργα γιατί οπωσδήποτε υποστηρίζουμε αυτή την πολιτική και βεβαίως αλλιώς δεν θα είχαμε και λόγο ύπαρξης. Τέλος για τον κύριο Μίτσελ να πω πως ε, Οπωσδήποτε παίρνουμε πολύ σοβαρά την έκκλησή του. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μέιστατ, ήταν στην Επιτροπή σας το Σεπτέμβριο και είναι διατεθειμένος να έρθει ανα πάσα στιγμή. Αν θέλετε λοιπόν να προετοιμάσουμε ένα έγγραφο για το πώς ε, φέραμε 50 δισεκατομμύρια περισσότερα δάνεια σε μικρομεσαίες ε, επενδύσεις και στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής σε περίοδο κρίσης, ευχαριστώ να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Κιούτας, θέλετε να απαντήσετε. Πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ συναδέλφους. Όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή τη συζήτηση είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχετε γύρει. Ακόμα και τα προβλήματα που ανέφεραν οι πράσινοι. Και εγώ περιμένω τις τροπολογίες σας για να έχουμε και μια βάση συζήτησης για περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σα υπενθυμίζω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία τροπολογιών είναι 7η Φεβρουαρίου. Θα εξεταστούν τροπολογίες 28 Φεβρουαρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 15 Μαρτίου και στην Ολομέλεια, μάλλον στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, γιατί γνωμοδοτούμε, 28 Φεβρουαρίου και όλα αυτά τα θέματα θα έρθουν στην Ολομέλεια τον Απρίλιο, την Ολομέλεια του Απριλίου. <coughs> Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία. Θα σας δώσω λίγα λεπτά για να ταξινομήσετε τα χαρτιά σας. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας. So I can't read it now. <laughs> <laughs> <laughs>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 Θέλω να ζητήσω κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω την κάρτα μου σήμερα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, όλοι αυτοί που είναι ένοχοι απώλειας και δεν έχουν τις κάρτες τους, λοιπόν, δύο από, το, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές χωρίς κάρτα. Κάποιος άλλος? Είμαστε όλοι έτοιμοι. Κύριε Κοζές, έχετε την κάρτα σας. That's all right. We can keep it. We can keep... Εντάξει, μπορούμε να κρατάμε λογαριασμό. Δύο μέλη του ΕΛΚ, ένα μέλος του ΕΛΚ και δύο από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές δεν έχουν κάρτα. Μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. δοκιμαστική ψηφοφορία. Πατήστε όποιο κουμπί θέλετε. Yep. Happy buttons Okay. We've got We haven't got everybody pressing their buttons yet. Δεν έχετε πατήσει όλοι το κουμπί σας. 37 είναι συνδεδεμένοι, 34 ψήφισαν, 35-38 συνδεδεμένοι με το σύστημα. 36, εντάξει. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση του κύριου Κούτας για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιωτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 1 ψήφι κατά αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεν μου αρέσει αυτός ο κατάλογος, ε, λέει πρόεδρος. Τροπολογία 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά ίσως, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω από τα χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε ήδη όλοι. Δύο ΕΛΚ και δύο συντηρητικοί δεν έχουν, δεν έχουν <laughs> κάρτες. Πέρας προφορίες. 28 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται επομένως. Τροπολογία 8. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 11 είναι σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 12, παρακαλώ. Άρχεται. Πέρας. Ισοψηφία. Κύριε Χαρκουμάκ, πώς ψηφίσατε. Έχουμε τέσσερις ακόμα που υπερψηφίζουν χωρίς κάρτα, εντάξει. Εγκρίνεται επομένω. 13 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C, λατινικό. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται και αυτό. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά, δεν βλέπω να σηκώνται πολλά χέρια, άρχεται ψηφοφορία στο δεύτερο τμήμα. Πέρας εγκρίνεται σαφώς. Συμβιβαστική ε ή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47, ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. 48 <clears throat> υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές κρίνεται συμβαστική F σίγματα ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε <clears throat> στην F σίγματα φελνικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται με τα τσαρούχια. Απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τις μεμονωμένες των τροπολογίες. Τροπολογία 50. Ψήφι υπέρ. <clears throat> Κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες οι υπόλοιπες εκπίπτουν και οι 59. Όλες, όλες. Συμβαστική τροπολογία Z, Ζ. λατινικό σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΙΤΑ, H, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία I, θ, ψήφι υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Τροπολογία J, συμβαστική Ι, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 76, υπέρ, κατά, δεκτή. 77, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική K, λατινικό, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85, υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 86, υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε για την 86, άρχεται ψηφοφορία. Δύο. Δύο ψηφίζουν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρόσθετοι. Είσαστε κατά εσείς από τη συντηρητική ομάδα. Τρεις κατά. Επομένως δεν γίνεται δεκτή. 87 ψήφοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία L, λατινικό υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 95 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχω διαφορετικές ενδείξεις από τον εισηγητή. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 ναι, ναι, <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ερέχουμε την 104. Ψηφίσατε όλοι. Δεν κρίνεται. Τι λένε αυτοί που δεν έχουν κάρτα. ή άκαρτοι. Α, κάρτα στάση εποχής. Εντάξει, εγκρίνεται. 105 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 106. Έλεγχος. Εντάξει, την 105. Άμα σηκώνετε τα χέρια σας είναι πολύ πιο εύκολο εξάλλου, λέει η 105 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. απορρίπτεται. 106 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συνδυαστική N υπέρ, κατά M αποχές δεκτή. 115 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά αποχές Νομίζω πως γίνεται δεκτή, αλλά να την επαληθεύσουμε την 116. Ψήφισαν όλοι. Δεκτή. Η επόμενη είναι η 124 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ. Έχει καταπέσει. 131 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 132 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος είναι μόνο το Ναι. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ούτως ή άλλως. 133 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 135 Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 136 υπέρ. Κατά. Ε. Άμα βλέπω τρία χέρια μόνο, πρέπει να επαληθεύσουμε. Λοιπόν, 136 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε την 139. Ψήφισαν όλοι. Δεκτή. Συμβιβαστική ομικρόν. Σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο μέρος 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική πι υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο παραγραφός 16 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 167 υπέρ κατά αποχές δεκτή 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Δεκτή. Μέρο τρίτο υπέρ κατά εποχέ δεκτό. 173 υπέρ κατά εποχέ δεκτή. 12 υπέρ. Όχι, κατά πίπτη. 174 υπέρ κατά. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αρχικό κείμενο παράγραφος 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε. Την 177. Ωραία άρχη τη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Επόμενες καταπίπτουν 181 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές δεκτή 184 υπέρ κατά αποχές δεκτή 185 υπέρ 185 υπέρ ε, σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ δεν, δεν μπορώ να μετρήσω τους συντονιστές δεν, δεν ψηφίζουν μαζί οι ομάδες. Λοιπόν, 185 υπέρ. Κατά. Ωραία, απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ. Α, όχι, είναι ίδια. 193 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά αποχές δεκτεί. Οι υπόλοιπε καταπίπτουν. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την 197. Πόσους πρέπει να προσθέσουμε τρεις. Οπότε απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 200 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 202 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Νομίζω, αλλά να επαληθεύσουμε τη 202. Ψήφισαν όλοι. Και τρεις κατά, οπότε απορρίπτεται. 203 υπέρ. Κατά αποχές. Και 203, ξανά παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά εποχές δεκτή να, επαληθε... Ε, να επαληθεύσουμε όμως γιατί ήταν τσίμα τσίμα νομίζω αλλάζεται συνέχεια μυαλό δεκτή 208 υπέρ κατά εποχές δεκτή 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 210 υπέρ κατά αποχές απορριπτείται 211 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Να το επαληθεύσουμε όμως το δεύτερο μέρος. Υπάρχει κάποιος άλλος να ψηφίσει. Πέρας. Δεκτή. Και ηλεκτρονική ψηφοφορία στην έκθεση όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και με άλλους τρεις υπέρ. Έχουμε 35 υπέρ, 6 κατά 4 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή.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 χρηματοπιστωτική ομίλη. Right, could we have quiet, please? Could we Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. <clears throat> Μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ώστε ο Θεόδωρος να παρουσιάσει την εκθεσή του. we, we do want to carry on with Ναι, να συνεχίσουμε σας παρακαλώ. Εξέταση της ε, εκθέσεως του κυρίου Θεόδωρου Στολογιάν για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Θεόδωρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το σχέδιο οδηγίας. Στόχος να βελτιωθεί η επιπλέον εποπτεία ομίλων, χρηματοπιστωτικών ομίλων. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν προτείνουν να πετύχουμε το στόχο αυτό σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση, αυτό που λέμε quick fix, οδηγιών που ήδη υπάρχουν για την συμπληρωματική εποπτεία και αυτό είναι και το αντικείμενο του σχεδίου της οδηγίας που προτείνει η Κομισιόν. Δεύτερο βήμα, μέχρι το τέλος του 2011, είναι η πιο θεμελιώδης μεταρρύθμιση από την Κομισιόν του θέματος αυτού και πιθανώς να έχουμε πρόταση της Κομισιόν του χρόνου. Η Κομισιόν βέβαια έκανε την πρόταση αυτή την πρώτη φάση, μας την έστειλε και το Συμβούλιο ήδη συμφώνησε για τις αλλαγές που επιβάλλονται για τις οδηγίες. Σήμερα έχουμε τις προτάσεις τροπολογιών, τις δικές μας, στο σχέδιο της Κομισιόν. Και οι τροπολογίες μας έχουν συντονιστεί κατά κάποιο τρόπο ήδη με τις τροπολογίες του, κοινο... του Συμβουλίου. Πριν επισημάνω τις πιο σημαντικές τροπολογίες, Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Ιβο Ιβάνε, σύμβολό μας στην Επιτροπή, που με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί γίνονται πολλές τεχνικές αλλαγές, προκειμένου να οι οδηγίες μεταξύ τους να μην χαρακτηρίζονται από ανακολουθία, σε σχέση με αυτό που απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Συν τις ειδικέ μας οδηγίες για, την ε, νέα, για τις νέες υποπτικές αρχές και ως προς την ορολογία και τον συσχετισμό όλων αυτών των νέων κανονισμών και οδηγιών. Τι κάναμε στην έκθεση αυτή. Πρώτον, έχουμε αλλαγές για την οδηγία όσον αφορά την φερικιότητα 2. Ε, για, τον ασφαλιστικό κλάδο και θα ισχύει μέχρι το 12 αυτό. Το Συμβούλιο επίσης για τροπολογίες και για την οδηγία Φεργιώτα 2. Άλλες τροπολογίες. Ε, αφορούν τις ευρωπαϊκές ε, υποπτικές αρχές. Όλες οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από αυτές τις αρχές θα γίνονται από την Κοινή Επιτροπή. Άλλες τροπολογίες έχουν στόχο τη διαφάνεια. Ιδιαίτερα υπάρχει μια τροπολογία σχετικά με τον κατάλογο και την δομή του δημοσιονομικού ομίλου που θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημοσίευσης. Σήμερα αυτός ο κατάλογος είναι μυστικός. Δεν δημοσιεύεται μέχρι στιγμής. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί και να δοθεί ορισμός τι εννοούμε με αυτές τις μικτές ε, εταιρείε holding δημοσιονομικού χαρακτήρα, ε, συγγνώμη, ε, χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, όπως επίσης και τους διαχειριστές των ταμείων, επενδυσιακών ταμείων. Επίσης έχουμε μια τροπολογία για να υπάρχουν τεστ κοπόσεως σε σχέση με κάθε χρηματοπιστωτικό όμιλο. Βέβαια, φυσικό είναι να υποθέσετε ότι υπάρχουν λόμπι τα οποία κινούνται σε σχέση με τα σχέδια αυτά τροπολογιών και ήδη έχω συναντήσει μερικούς εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τράπεζες, ασφάλειες. Γενικά συμφωνούν με την πρόταση της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Υπάρχει μια επιφύλαξη όσον αφορά τα τεστ του κοπόσεως. Κυρίως ε, η του ασφαλιστικού κλάδου μου είπανε να προσέχουμε μην τυχόν δημιουργήσουμε ε, διάφορα επίπεδα με διαφορετικούς κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή μια ασφαλιστική εταιρεία που ανήκει σε έναν όμιλο, χρηματοδοτικό όμιλο, να υποστεί και αυτή το τεστ κόπωσης, ενώ μια άλλη εταιρεία ασφαλιστική που δεν πληρεί, ας το πούμε, ε, τους όρους, το όριο μάλλον, το κατόφι να μην συμπεριλαμβάνεται στο τεστ κόπωση. Αυτές είναι οι κύριες αντιρρήσεις που άκουσα μέχρι στιγμής. Βέβαια θα έχω και άλλες συναντήσεις για το σχέδιο οδηγίας. Αυτά είχα να πω. Αυτές είναι οι κύριες αλλαγές που προτείνουμε. Θα ακούσω τα σχόλιά σας, τις τροπολογίες σας και θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση μετά με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε συμβασμό. Αν και δεν υπάρχουν πολλές τροπολογίες στη δική μας έκθεση που διαφέρουν πολύ από τις τροπολογίες Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πίτερ Σκίνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω τις τροπολογίες του εισηγητή και θέλω να επενέσω το έργο του, το οποίο φυσικά έγινε μαζί με και σκιώδεις εισηγητές και την, ε, τα άλλα μέλη της Επιτροπής, η προσπάθεια να λησαβονοποιηθεί η οδηγία Φερεγγιότητος 2. Και σε άλλες οδηγίες βέβαια ήταν απαραίτητες ε, αλλαγές. Εμείς δεν θα καταθέσουμε τροπολογίες τώρα σε αυτή την ε, έκθεση, ενώ δεν συμφωνούμε για τα πάντα και δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, νομίζουμε ότι είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Είναι πολύ χρήσιμη συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Είναι πολύ θετικό και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλό αποτέλεσμα. <clears throat> Ίσως οι τροπολογίες σας μπορεί να χρειαστούν κάποιες μικρές τροποποίησεις και ποια είναι τα θέματα τα οποία αξίζουν περισσότερη συζήτηση. Χαιρετίζω παραγωγικά χάρη την τροπολογία 31 η οποία ζητά από τη Μικτή Επιτροπή να παρακολουθήσει όλες τις ρυθμιζόμενες ε, οντότητες που είναι τμήμα του χρηματοπιστωτικού μήλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις τρεις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές πρέπει να συνδέονται όμως αυτές οι οντότητες και με τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με πιστοδοτική και ασφαλιστική δραστηριότητα. Η δημιουργία περαιτέρω φορέων όμως από την Κομισιόν αυτό είναι κάτι που αξίζει να το εξετάσουμε. Κάποια θέματα είναι πρόσθετα αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα νέο επίπεδο ρυθμίσεων. Έχουμε ουσιαστικά τους ίδιους ρυθμιστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες εταιρείε. Νομίζω ότι είναι μια πρόσθετη και περιττή περιπλοκή. <clears throat> να υποχρεώσουμε τη δημιουργία αυτών των νέων φορέων. Ουσιαστικά είναι πολύ λίγοι άνθρωποι, είναι πολύ λίγοι υπόλοιποι που έχουν στη διάθεσή τους. Νομίζω ότι αυτό θα συμπαρασύρει πάρα πολύ περιτές περιπλοκές. Έχω κάποιες ανησυχίε σε σχέση με τις εξουσίες οι οποίε προτείνονται από τον εισηγητή για την ε, μεικτή επιτροπή. <clears throat> Εγώ θέλω το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει τα σωστά επίπεδα και να διευρύνει τις εξουσίες μεικτής επιτροπής. Έχω δύο ανησυχίες. Καταρχήν, αν μπορεί κανεί να δώσει στη μεικτή επιτροπή μια νομική προσωπικότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό και γι' αυτό η τροπολογία 23 που σας ζητώ να την επανεξετάσετε κύριε Σιγητά του να γίνουν αυτές οι <clears throat> αρμόδιες αρχές αυτή η ορολογία που, είναι, που δίνει μια νομική προσωπικότητα δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη. Πρέπει να διευκρινίσουμε το ρόλο των ε, φορέων εποπτείας αλλά δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να εφεύρουμε νομικές αρμοδιότητες για αυτές τις επιτροπές και επίσης για την, το τεστ τροπολογία 39 που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Ίσως υπάρχει πολύ διακριτική ευχέρεια της ε, Μικρής Επιτροπής εδώ. Εγώ θα ήθελα ο ρόλος της να είναι πιο σαφής και να καθορίσουμε τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Να δούμε αν είναι γεμάτο ή άδειο το ποτήρι σε αυτή την περίπτωση. Αν περιμένουμε κάποιοι άλλοι φορείς να καλύψουν αυτό το ρόλο, μπορεί να περιμένουμε για πάρα πολύ καιρό. Αλλά για τη δημοσιοποίηση των τεστ κοπόσεων στις ιστοσελίδες, αυτό μπορεί να γίνει και με δράση του τοπικού ρυθμιστή. Και επίσης, <clears throat> τι θα γίνει με την περίπτωση όπου υπάρχει ε, μια σειρά συναλλαγών σε επίπεδο εκτός αγορών <clears throat> για τις τράπεζες και τους χρηματοοικονομικούς φορείς. Δηλαδή σε ποιο βαθμό θα πρέπει να εμπλέκεται το ενεργητικό του σε τέτοιου είδους συναλλαγές και ίσως μπορούμε να ακολουθήσουμε λιγάκι το αμερικανικό μοντέλο και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά επί τη βάση του τι ακριβώς μπορούν να γίνουν σε αυτό το τομέα επί τη βάση της αμερικανικής εμπειρίας. Και επίσης μπορούμε να δούμε και τη, σταθερότητα, την χρηματοοικονομική σταθερότητα και ενδεχομένω η τροπολογία σας 52 μπορεί να επεκταθεί <clears throat> τους ε, ομίλους να επενδύουν πάνω από 3% του κεφαλαίου τους επίπεδου 1 σε τέτοιες μορφές εναλλακτικών επενδύσεων. Όχι όλο το κεφάλαιο, αλλά 3% του κεφαλαίου tier 1, δηλαδή επίπεδου 1, σύμφωνα με τη Βασιλεία 2. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτή την επόμενη φορά και θα είμαι έτοιμο να ακούσω αυτά που έχει να πει ο εισηγητή. Okay, Uh, right. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι σκιώδη εισηγήτρια από του φιλελεύθερου. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Μπορώ να συμφωνήσω γενικά με πολλά από αυτά τα οποία ελέγχθησαν και με την θέση του εισηγητή. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν τα τεστ κοπόσεως ώστε να καλυφθούν τα κενά ρύθμισης. Και νομίζω ότι η κοινή επιτροπή, η μεικτή επιτροπή θα πρέπει να έχει τρόπο να παρακολουθεί αυτά τα γεγονότα και μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια πλήρης κάλυψη χωρίς να υπάρχει επικάλυψη και σε μερικούς χώρους και κενό σε άλλους χώρους. Θέλω λοιπόν να επαληθεύσουμε και πάλι ότι έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε μια πλήρη κάλυψη και αυτός χωρίς επικαλύψεις και αυτός είναι ο στόχος των τροπολογιών. Και εγώ κάπως ε, νιώθω σύγχυση σε σχέση με το πόσους περισσότερους φορείς και επιτροπές χρειαζόμαστε για την υποπτία. Μήπως παίρνουμε κάτι μπερδεμένο και το κάνουμε ακόμα πιο μπερδεμένο. <clears throat> Θα ήθελα λοιπόν να ελεγχθεί αυτό και πάλι χαιρετίζω το γεγονός ότι η, εποπτική αρχή για τα αξιόγραφα περιλαμβάνεται σε αυτή τη ρύθμιση και δεν την αφήνουμε από <clears throat> στην άκρη. Και εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο έχει να κάνει με την, ε, με την νομική προσωπικότητα των εποπτικών επιτροπών. Έχουν μεγάλο πρόβλημα ανθρωπίνου δυναμικού και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συντονίζουν. Αλλά αν μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι κατάλληλοι πόροι πηγαίνουν στη σωστή μορφή εποπτείας, αυτό είναι κάτι το οποίο εμπίπτει στην εμβέλεια του κανονισμού της οδηγίας καλύτερα. Ναι, μπορεί να πρέπει να διευρυνθεί το φορέας αυτός και να έχει περισσότερους, περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά δεν πρέπει να το πνίξουμε με το να το επιφορτήσουμε το σώμα αυτό με αρμοδιότητες τις οποίες δεν τις έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το σώμα και σιγά σιγά θα πρέπει να το βοηθήσουμε να μεγαλώσει χωρίς να το υπερφορτώσουμε. Αυτά λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα καταθέσουμε πάρα πολλές τροπολογίες, απλώς θέλουμε να ελέγξουμε ότι έχουμε καλύψει τα κένα και τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν. Ο Φίλιπ Λάμπερτς τώρα έχει το λόγο. Για την ε, επειδή οι δύο προηγούμενοι ομιλητέ είναι υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμοσύνη, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Συμφωνώ και ευχαριστώ τον εισηγητή επίση. Ιδιαίτερα για την έκθεση. Εμεί δεν έχουμε επιμέρου τροπολογίε. Η μία, μία τροπολογία έχουμε μόνο που μα ενδιαφέρει. Ξέρουμε ότι η οδηγία αυτή ε, αφορά τις διάφορε οντότητε. υπάρχουν ειδικού τύπου οχήματα στον χώρο αυτό που δεν πρέπει να ρυθμίζονται. Που να έχουν δηλαδή να είναι ιονοί όμιλοι. Σε αυτό μόνο χρειαζόμαστε μια διευκρίνηση. Με αυτή την εξαίρεση συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ανάφεραν ήδη οι δύο συνάδελφοι και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σίγουρα θα πετύχουμε συμφωνία. Η Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Η αρχική έκθεση της Κομισιόν ήταν αρκετά καλή και η έκθεση του εισηγητή φυσικά σωστά στηρίζεται σε αυτό. Περισσότερο μια ερώτηση έχω να κάνω. Γιατί το IFM δεν μπήκε στο αρχικό κείμενο της Κομισιόν υπήρχε λόγος. Αν έμπαινε μέσα στο κείμενο, τι επίπτωση θα είχε, δηλαδή πόσες εταιρείε των ομίλων θα επηρεάζονταν από αυτό, αν γινόταν μια μελέτη αξιολόγησης. Γιατί έγινε αυτή η παράληψη, είναι σκεμμένη. Δεν ξέρω αν κάποιος από την Κομισιόν θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Λοιπόν, θα συμφωνούσα να μπει το IFM άμα σε εξηγηθεί γιατί δεν μπήκε στην αρχή, από την αρχή μάλλον. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έχουμε ένα εκπρόσωπο της Κομισιόν. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν συμπεριλήφθηκε το, το IFM. Ναι, η πρόταση δεν, ε, όταν δημοσιευθήκε η πρόταση τον Ιούνιο δεν είχε υπάρξει ακόμα, δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το IFM εκείνη την εποχή. Τώρα φυσικά είναι δημοσιευμένη η δημιουργία του, ήταν απλώς, απλώς τεχνικός ο λόγος που δεν το λάβαμε υπόψη μας. Εγώ πιστεύω και εγώ ότι το AIFM θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην περίπτωση αυτή. Δεν θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Εισηγητά, <clears throat> για να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και είμαι φυσικά έτοιμος να συνεργαστώ με τους οι εισηγητές και τους ε, υπόλοιπους ενδιαφερεμένους και στη συνέχεια μπορούμε να ετοιμαστούμε να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν η προθεσμία τροπολογιών. Είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου, εξέταση τροπολογιών στις 28 Φεβρουαρίου. 21 Μαρτίου θα ψηφίσουμε ώστε να έρθουμε στην Ολομέλεια του Μαΐου. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και περνάμε στο σημείο 14 συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων με εισηγητή τον Πίτερ Σκίνερ. Σύντομα θα είμαι, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, πιστεύω ότι η εγγύηση των ασφαλίσεων θα είναι από κάθε άποψη ένα πολύπλοκο θέμα. Και ουσιαστικά έχουμε μια πολυπληθώρα προσεγγίσεων από τα κράτη-μέλη και τώρα που μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της προστασίας των φορολογουμένων, βλέπουμε ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια ενέργεια. Νομίζω ότι η αλληλεπίδραση με το Solvency 2, φεραγκαιότητα 2, που είναι και αυτό ένα νομοθέτημα προστασία των καταναλωτών, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε και την προσέγγιση που έχει ακολουθηθεί στον τομέα του τραπεζικό. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι <clears throat> ότι οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν είναι τράπεζε και οι τράπεζε δεν είναι ασφαλιστικέ εταιρείε. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποίηση μεταξύ των δύο και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει επακριβή και εκπεφρασμένος διαχωρισμό. Ξέραμε στην περίπτωση του Solvency 2 να ξέρουμε ότι η ασφάλιση των η εγγύηση των ασφαλίσεων θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί στη συνέχεια. Εγώ θα ήθελα κάποιος να μου πει αν έχουμε το IGS γιατί δεν πρέπει να έχουμε και υποστήριξη των ομίλων, των ομάδων μάλλον καταναλωτών. Όταν το χρειάζονται αυτό λοιπόν οι καταναλωτές, το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και να επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην κίνηση τέτοιων κεφαλαίων. Εγώ δεν νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο τελικό επίπεδο, είμαστε απλώς στο επίπεδο συμπληρώσης των κενών στο μοσαϊκό αυτό. <clears throat> Επομένως, δεν έχουν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοια συστήματα, αλλά οι μεγαλύτερες χώρες έχουν ένα τέτοιο σύστημα και το Solvency 2 <clears throat> δείχνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πολλά θέματα σε επίπεδο εθνικών συστημάτων εγγύησεων Κατά την άποψή μου λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια αρχή ότι η κάθε χώρα ακολουθεί το δικό της σύστημα και όχι μια ενοποιημένη αντιμετώπιση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πούμε επίσης ότι όταν πτωχεύει ένας ε, εγγυητής ασφαλίσεων δεν έχουμε την ίδια κατάσταση όπως με τις ε, τράπεζες αλλά οι τοπικοί ρυθμιστές θα πρέπει να υπομισθούν την ε, ευθύνη για τέτοιου είδου πτωχεύσει, πολύ περισσότερο από τις, τραπέ... οι οποίες μπορούν να πτωχεύσουν ανα πάσα στιγμή όπως έχουμε δει πρόσφατα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και μεγαλύτερη δυνατότητα διαμεθοριακής λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιριών αυτών που δημιουργούνται με διάφορες, ε, διάφορα ονόματα σε διάφορες χώρες έχουν ε, θηγατρικές και υποκαταστήματα περισσότερο υποκαταστήματα βέβαια λόγω της ε, κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Επομένως μπορεί να αγοράσουν κάποιοι από χώρες, σε χώρες και από εταιρείε που δεν ξέρουν πραγματικά ποιος είναι ο ρυθμιστής της μετρικής εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προστασία μετά από την ε, έρευνα που κάναμε για την Equitable Life. Βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν και χρειάζεται να διατηρήσουμε την κριτική στάση που έχουμε σε σχέση με εταιρείε οι οποίε δεν λειτουργήσαν σωστά. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την αρχή της χώρας προέλευσης, μπορούμε να εξασφαλίσουμε περίπου 100% πρόσβαση στο σύστημα εγγύησεων παράλληλα με άλλα συστήματα εγγύησεων. Και εγώ νομίζω ότι όλες οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σεβαστές. Έχουμε στοιχεία ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν καταρρεύσει με ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος ήταν ναι, υπήρξαν κάποιες εταιρείε οι οποίες απέτυχαν σε κάποιο επίπεδο, αλλά δεν είχαμε τέτοιου είδου καταστροφικές καταρρεύσεις όπως σε άλλους τομείς και εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε κάποιες ε, διαδικασίες τροχοπέδησης των προβλημάτων αυτών. Νομίζω ότι η ΑΕΟΠΑ θα πρέπει να εμπλακεί όπως και η AGS για να δημιουργήσει δεσμευτικά πρότυπα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε ίσως στην οδηγία Omnibus 2. Αλλά επειδή δεν υπάρχει ακόμα ένας ε, νομικός ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ έχω προβλήματα όταν ζητείται το σύστημα IGS των εγγυήσεων να καλύπτει τέτοιου είδους νομικά πρόσωπα. Εάν δεν έχουμε τέτοιο ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και σε σχέση με τη μορφή του IGS, η Κομισιόν υπερθέλει ένα ταμείο ex ante, Αυτό ίσως ε, το κάνει λόγω αυτών που συνέβησαν στον τραπεζικό τομέα, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν οι ίδιες συνέπειες στον τομέα των ασφαλίσεων. Όπως σας είπα, δεν υπήρξαν τέτοιου είδους καταρρεύσεις ασφαλιστικών εταιριών και <clears throat> μπορεί κάποιος να μπει σε ένα σύστημα ασφάλισης από το οποίο δεν μπορεί να βγει, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα σαν μια κατάρρευση τραπεζών. Η χρηματοδότηση εξάντε λοιπόν θα δημιουργήσει προβλήματα. Το να δίνουμε λοιπόν υποχρέωση αυτού του είδους για εξάντε ταμεία δεν είναι πρόσφορο στην περίπτωση αυτή γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν καταραίουν μαζικά, πολύ σπάνια καταραίουν και εξάλλου έχουμε ένα, μια πληθώρα εθνικών συστημάτων εγγύησης. Με το να έχουμε ένα ενιαίο μοντέλο μονάχα αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όταν ήδη έχουμε λόγω πολλών αλλορυθμίσεων αρκετή ε, ανακατοσούρα στις αγορές και στις εταιρείε. Ξέρει η Κομισιόν ότι έχουμε στην Οδηγία 2 σημαντικές κεφαλουχικές απαιτήσεις. Και επίσης απαιτείται και ένα μικρό αποθεματικό πέραν των κεφαλουχικών ε, απαιτήσεων. Και έχουμε και τις εταιρείε πιστοληπτικής αξιολόγησης οι οποίες κάνουν και αυτές τη δική τους αξιολόγηση και ζητούν περαιτέρω κεφάλαιο. Λοιπόν, πόσο κεφάλαιο πρέπει να έχει κανείς, άμα αρχίσουμε και ξεπερνάμε ε, κάποια όρια ασφαλείας, θα υπάρχει αυτόματη αίτηση για περαιτέρω κεφάλαιο. Επομένως, μια εξάντεκτον εκ των προτέρων αίτηση για δημιουργία ταμείων ασφαλείας δεν ευσταθεί. Αυτά είναι τα στιγμή τα οποία ήθελα να σας αναφέρω. Uh, ο e κύριος Καράς από το ΕΛΚ δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ ο οποίος θέλει να τον αντικαταστήσει. κυρία Λούλινγκ δεν είπε ότι θέλει να λάβει. Ο κύριος Σμιτ, Όλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο αυτό. Πάνω κάτω συμφωνώ με τον Πίτερ. Οι εξηγήσει στη Λευκή Βίβλο της, ε, της Κομισιόν δεν με πείθουν για πολύ ότι είναι σωστές όπως μας υποβάλλονται αλλά ο Πίτερ είναι ο εμπειρογνώμονας. Εγώ είμαι υπεύθυνο για, για την έκθεση σχετικά με τι αποζημιώσει και υπάρχουν ορισμένε ομοιότητε. Δεν ξέρω αν για αυτή εδώ τη λευκή βίβλο, αν αυτό θα έπρεπε να γίνει και για τι ασφαλίσει. Γιατί οι ασφαλίσει είναι άλλο πράγμα, όπω είπε και ο Πίτερ. Η προστασία του καταναλωτή είναι το υπαριθμό 1 για την Κομισιόν καλύπτεται από τη Φεραγγιότητα 2. Ναι, όπως είπε ο Πίτερ. Βέβαια, οι ερωτήσεις μου μάλλον δεν αφορούν τον εισηγητή, αφορούν περισσότερο την Κομισιόν. Θέματα ανταγωνισμού. Καλύπτεται από τη Λευκή Βίβλο. ούτε και γι' αυτό είμαι πολύ πεπισμένο. Η, η δημοσιονομική σταθερότητα. Υπάρχουν θέματα που αφορούν την, ε, ε, τις ασφαλίσεις σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Γιατί δεν είχαμε και πολλές πτωχεύσεις στον κλάδο αυτό. Αν λειτουργεί σωστά η ενιαία αγορά, θα έχουμε οπωσδήποτε διασυνοριακά προβλήματα και θέματα. Και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά είναι το σύστημα προχρηματοδότησης. Νομίζω η πλειοψηφία της Επιτροπής συμφώνησε ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, τι ζητάμε από το χρηματοπιστωτικό κλάδο, τις τράπεζες κλπ. να ξέρουν τι έχουν να πληρώσουν. Γιατί αν δεν πληρώσουν αυτοί θα πληρώσουν οι καταναλωτές. Ή μάλλον ό,τι επιβάλλουμε σε αυτούς να πληρώσουν θα το πληρώσει τελικά ο πελάτης ή ο καταναλωτής. Όλα αυτά τα υποβάλλω περισσότερο με τη μορφή ερωτημάτων. Και νομίζω πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά στην Επιτροπή μας και μεταξύ των σκιωδών εισηγητών των ομάδων. Και θα ακούσω με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση της Κομισιόν. Γιατί θα πρέπει να πιστώ με καλύτερα επιχειρήματα υπέρ των προτάσεων αυτών. Αυτά είναι τα δικά μου συμπεράσματα. Η Βίκη Σας ευχαριστώ που προχωρείτε τόσο γρήγορα. Συγγνώμη, έχασα την αρχή της ομιλίας του εισηγητή. Καλό είναι να τρέχω πιο γρήγορα στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου ίσως. Νιώθω κάποια σύγχυση σε σχέση με το σύνολο αυτό θέμα των εγγυήσεων για τις ασφαλίσεις. Είναι τόσο διαφορετικές οι ασφαλίσεις από τον τραπεζικό τομέα. Ξέρετε, δεν σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά. Οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν είναι τράπεζε, δεν έχουν τεράστια έκθεση η μία στην άλλη. Οπότε ο κίνδυνος είναι να χρεοκοπήσουν οι... ταυτόχρονα κάποιες ασφαλιστικές εταιρείε. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τους κινδύνου στον τραπεζικό τομέα και για μένα αυτό είναι ο βασικό λόγο για τον οποίο ένα τεράστιο ταμείο εξάντε δεν χρειάζεται γιατί λόγω των συνθήκων ε, στη, στον ασφαλιστικό κλάδο. Σε αντίθεση με τις αντασφάλειες, οι οποίες συμφωνώ ότι είναι διαφορετικές, αλλά τις βασικές ασφάλειες ζωής, ε, ε, αυτοκινήτου κτλ. είναι διαφορετικές εταιρείε χωριστές, οι οποίες αν έχουν κεφαλιακή επάρκεια μέσω της οδηγίας φερεγκαιότητα 2 θα προστατεύονται. Βεβαίω δεν μπορούμε ποτέ να αποτρέψουμε τη χρεοκοπία μια εταιρεία ποτέ. Αυτό έχει συμβεί. Γι' αυτό ο καταναλωτή χρειάζεται προστασία. Κάποια είδου εγγύηση. Για το κάθε κράτο μέλο το βλέπει διαφορετικά. Άλλα έχουν, άλλα δεν έχουν. Και αντιλαμβάνομαι πω αυτό βεβαίω μπορεί να μπερδεύει του καταναλωτέ όταν εξετάζουν προϊόντα που του προσφέρονται από διαφορετικές εταιρείες βασίζονται σε διαφορετικά κράτη-μέλη η πρόταση ότι χρειαζόμαστε πλήρως εναρμονισμένο σύστημα για να ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα και αυτό νομίζω παραπάει. Νομίζω πως οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν τις εκθέσεις, διαφορές στα διαφορετικά συστήματα, οπότε υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, τώρα δεν νομίζω ότι να χρειαζόμαστε κανένα ταμείο, ένα ταμείο το οποίο από ό,τι κατάλαβα πληρώνουν ε, οι εταιρείε, ε, αλλά νομίζω το καλύτερο το οποίο θα ήταν ήταν κάτι το οποίο θα πληρώνουν ad hoc εταιρείε και μετά θα πληρώνονται από αυτό όταν θα υποβάλουν κάποιο αίτημα. Αυτό νομίζω είναι το λογικότερο. Οπότε όπως είπα δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε πλήρη εναρμόνιση σε αυτό το επίπεδο ούτε κάποια μαζική προχρηματοδότηση. Ένα ερώτημα από την αξιολόγηση, αξιολό, αξιολόγηση επιπτώσεων της δεν είχαν εξετάσει την ε, ε, ασφάλιση αυτοκινήτων, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να εξεταστεί όπως είπα και ούτε και ασφάλιση ζωής ούτε τίποτα, οπότε δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Οπότε σε αυτά θα μείνω ευχαριστώ. Αστρίτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Δεν είμαι. Αυτοί που ορίζονται θα πρέπει να είναι παρόντες όταν συζητιέται η έκθεσή τους. Είναι θέμα αρχής για μένα. Επίσης σας ομολογώ, επειδή είχα άλλες δουλειές, ακόμα δεν είχα την ευκαιρία να μελετήσω αυτό το σχέδιο έκθεσης. Έχω όμως μία πρωτόγονη ερώτηση προς τον εισηγητή. Έχουμε τη φερεγγιότητα 2. Έχουμε τι νέες δομές εποπτείας των ασφαλίσεων. Δεν αρκεί αυτό. Ευχαριστώ πρέπει να εξηγήσω ξανά πως ο κύριος Κάρας έπρεπε να κάνει μια παρουσίαση στην εταιρική διακυβέρνηση στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και συμπίπτει. Γι' αυτό λείπει, αλλά είναι εδώ πέρα βοηθός του και κρατάει σημειώσεις. Οπότε θα είναι ενήμερος. Θα βάλω και τον εαυτό μου στον κατάλογο των αγορητών, μια που υπάρχει χρόνος, εγώ και ο Πίτερ συμφωνούμε σε κάποια πράγματα για την οδηγία Φερικαιότητας 2. Τέσσερα. Είχα κάποια πράγματα να πω, μπορώ να περιμένω για άλλη στιγμή, αλλά στην οδηγία είχαμε πει πως περιμέναμε κάποιο σύστημα εγγυήσεων και ζητήσαμε από την Κομισιό να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα στη διαβούλευση μετά την οδηγία είχα πει κάποια πράγματα και προσπαθώ να τα θυμηθώ αλλά αυτό το οποίο με δίδαξε κάποια πράγματα εμένα είναι το πόσο μεγάλη αντίσταση υπήρχε από κάποια κράτη-μέλη, κάτι το οποίο με εξέπληξε, αλλά μετά βίωσε όταν το εξέτασα είχαν κάτι που ισοδυναμούσε με κάποιο είδος εγγύησης. Απλά δεν ήθελαν κάποιο σύστημα το οποίο θα χρηματοδοτούνταν εκ των προτέρων και να πηγαίνουν περισσότερα λεφτά σε περισσότερα μέρη. Και πρέπει να το δουν πολύ προσεκτικά γιατί διαφέρει η ασφάλεια, η ασφάλιση από κράτος σε κράτος και οι εγγυήσεις πρέπει να είναι πλέον τελευταία λύση και έχουμε τόση προστασία των καταναλωτών που όχι μόνο είναι πολύ ακριβή αλλά δεν θα σκέφτεται και ο καταναλωτής και είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να γίνει αυτό. Και επιπλέον η πίεση θα υπάρχει πάντα να γίνεται μια πάρα πολύ γρήγορη πληρωμή από τα ταμεία εγγυήσεων αντί να υπάρχει κάποια υπομονή μέχρι να εκταμιευτούν τα λεφτά και υπάρχει και κάποια εκπαίδευση για να αντιληφθεί ο κόσμος πως δεν είναι όλα τα πράγματα στιγμία. Δεν είναι τα πράγματα ίδια με τον τραπεζικό τομέα όπου μπορεί κάποιος να καλέψει πως δεν μπορεί πλέον να κάνει τις πληρωμές του, δεν μπορεί να ζήσει και γίνει καμιά καταστροφή και σου καταστρέφει τη ζωή. Με την ποικιλία των ασφαλιών ε, ίσως να υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους μπορούμε να πούμε ναι, κάποιο, κάτι είναι πιο επίγον από κάτι άλλο. Οπότε, όπως και άλλοι, έτσι, και εγώ δεν είμαι υπέρ μιας ενιαίας λύσης ε, τυποποιημένης και να έχουμε ένα έτοιμο ταμείο έτοιμο να πληρώσει πρέπει να μπορούμε να το προσαρμόσουμε, αλλά γνωρίζω πως την ε, φερεγγιότητα 2, την οδηγία, το είχαμε ζητήσει, οπότε δεν ξέρω. Ασκούμε κριτική στην Κομισιόν για κάτι το οποίο ίσως ε, να μην είναι τόσο προχρηματοδοτούμενο σε πρόταση αυτή. Έχω κάποιους ομιλητές στον κατάλογο. Ο εισηγητή θα ήθελε να ακούσει την Κομισιόν, νομίζω, αν υπάρχει παρέμβαση. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν, ναι. Έχετε το λόγο. Κυρία Βολφ Λίντα. Thank you. Thank you for uh, the rapporteur, Peter. Κύριος Βολφ Λίντεν. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον Πίτερ, και ως παρενέβησαν συζήτηση. Κοιτάξτε, εμείς ε, προτείνουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση καθώς γνωρίζουμε τις εθνικές διαφορές των συστημάτων. Γύρω στις 12 χώρες έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Έχουμε δει προβλήματα εφαρμογής όταν τα συστήματα αυτά αντιμετωπίζουν πελάτες από διαφορετικές χώρες. Έχουμε δει αντίκτυπο της κρίσης και όπως βλέπετε Στη Λευκή Βίβλο αναφέραμε κάπως τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αυτό το σύστημα. Αντλήσαμε κάποια διδάγματα από την κρίση και όπως είπατε η φερεγγιότητα 2 δεν θα δημιουργήσει ένα σύστημα χωρίς αποτυχίες. Θα αυξηθούν πιθανότατα οι διασυνοριακές δραστηριότητες και θα μπορούσαμε να έχουμε και άνισους όρους ανταγωνισμού για χώρες από για εταιρείε από διαφορετικέ χώρε και ίσω να υπάρχει και κάποιο αντίκτυπο στι χρηματαγορέ. Αυτό το οποίο προτείνουμε, όπω είπα, είναι ένα ελάχιστο σύστημα. Στη Λευκή Βιβλία έχουμε αναφέρει κάποιες, τομεί τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Ξέρουμε πως πρέπει να υπάρχει η ουσιαστική ελευθερία των κρατών μελών να προσαρμοστούν στις παραδόσεις που έχουν και βεβαίως είμαστε από τις τελικές φάσεις, στην τελική φάση ανάλυση των σχολείων που έχουμε λάβει και βεβαίως θα επανέλθουμε με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Και αναμένουμε βεβαίως τη συνέχεια αυτής της συζήτησης και θα σας δώσουμε λοιπόν, λεπτομέρειες ή πληροφορίες που χρειάζεστε για το θέμα της ασφάλισης οχημάτων αυτό εξαιρείται από την πρόταση αυτή γιατί αντιμετωπίζεται σε άλλες οδηγίες. Αλλά όπως είπα, ευχαρίστως να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειάζεται για τις προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Αλλά κατά βάση στόχο έχουμε να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη τα σχόλιά σας. Μάλιστα. Πίτερ, έχεις πάλι το λόγο. Θα απαντήσω και εγώ για μερικές από τις παρατήρησεις που έγιναν. Η Βίκη αναφέρθηκε στα θέματα επανασφάλισης, αλλά η επανασφάλιση δεν έχει να κάνει παρά μόνο με επιχειρήσεις, δεν έχει να κάνει με καταναλωτές, είναι απλώς business to business. Θέλω να επανέλθω στο ρόλο της ίσης, όπως είπε η εκπρόσωπος του ΕΛΚ, η οποία τα καταφέρνει τόσο καλά, παρά το γεγονός ότι έχει να αντιμετωπίσει τόσες πολλές εκθέσεις. Ναι, είναι καλό να έχουμε το σύστημα ίσης, είναι καλό το ότι έχουμε τη φερεγγιότητα 2. Αυτά δεν εγγυώνται όμως μία απόλυτη έλλειψη πτωχεύσεων. <laughs> Είναι 99,9. Δεν υπάρχει εκτός από το σύστημα ασφάλιση, ε, των ε, ασφάλισεων, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα. Όπως είδαμε στην περίπτωση της Equitable Life, πρέπει να έχουμε μια συνεκτική αντιμετώπιση. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια ελάχιστη εναρμόνιση με την Κομισιόν. Αν θέλετε κάτι, ένα σύστημα που βασίζεται από σε ένα προηγούμενο ταμείο στο οποίο καταβάλλονται εγγύησεις, αυτό σημαίνει πλήρης ε, εναρμόνισης. Επίσης, πρέπει να καλύψουμε τα θέματα και των φυσικών προσώπων και των προσώπων νομικού, ε, νομικού χαρακτήρα των νομικών προσώπων. Ίσως η Μικτή Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε μια γενική συνεκτική αντιμετώπιση σε όλο το ευρωδαφός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγώ διαμφισβητώ τη λογική για το ταμείο αυτό. Όταν λέμε ότι υπάρχει πιθανότητα μονάχα μισό τα εκατό κάθε χρόνο να υπάρχει μια πτώχευση, αυτό σημαίνει ότι κάπου τα παρακάνουμε. Δηλαδή φοράμε ζώνη, φοράμε ε, τυράντες και έχουμε και κάποιον να κρατάει το πατελόνι μας να μην πέσει. Είναι υπερβολικό αυτό. Σας ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Θα σας υπενθυμίσω την ε, προθεσμία για τις τροπολογίες. 28 Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε την έκθεση αυτή. Έρχεται ένα μήνα, Πίτερ, για να τελειώσετε αυτή την έκθεση. 11 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, 11 Απριλίου στην Επιτροπή μας, ψηφοφορία το Μάιο, τον Ιούνιο στην Ολομέλη. Αυτό είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα στα διάφορα. Μπορώ να σας πω πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίασή μας. 3η 1η Φεβρουαρίου 9 με 12.30 και 3 με 6.30 έχουμε τελειώσει λοιπόν την συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ συνάδελφοι.